So, colleagues, even if in the dark, and uh, maybe we can start our meeting. First, I would like to have the agenda adopted, unless there are. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Είμαστε σκοτεινά, αλλά να ξεκινήσουμε. Ε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έχω μερικές ανακοινώσεις να κάνω. Θα ξέρετε ότι η συνεδρίασή μας στις 4 και 45 θα ακολουθηθεί από μια συνεδρίαση κοινή με την Επιτροπή Προπολογισμών για το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων. Οπότε να ξέρετε ότι οι καρτέλες με τα ονόματα είναι ήδη στις θέσεις για την κοινή συνεδρίαση. Επίσης, ο Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Μισελ Σαπά, και οι συνεργάτες του ε, επιβεβαίωσαν ότι θα παραστεί στον οικονομικό διάλογο με την ε, μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ στις 7 Μαΐου. Θα μας τιμήσουμε την παρουσία του λοιπόν ο κύριος Σαπά. Καλή είδηση για τους εξελισσόμενους τριμερείς διαλόγους, για την διατησία των εξασφαλίσεων, των αντασφαλίσεων. Ο τελευταίος γύρος ε, έγινε τον Απρίλιο των συζητήσεων με το πεδίο και τις εξαιρέσεις και προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το ΕΛΚ έκανε μια πρόταση προς το Συμβούλιο για να αποδειχτεί το σύστημα του Κοινοβουλίου για τις εξαιρέσεις, αλλά με αντάλλαγμα την ε, κατοπικοπή μέθοδο υπολογισμού του Κοινοβουλίου. Ε, πετεύχθη συμφωνία. Ο τριμερή διάλογο ολοκληρώθηκε πριν το προβλεπο... την προβλεπόμενη ώρα του ε, προγράμματο. Οπότε ο επόμενο γύρο ε, προβλέπεται στι 11 Μαου και εκεί ελπίζουμε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Επίση, ο τριμερή διάλογο για την οδηγία υπηρεσιών πληρωμή 16 Απριλίου. Τρίτο γύρο. Η Προεδρία υπέβαλε ένα συμβαστικό πακέτο για τους ε, ασφαλιστές και τα τρίτα μέρη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τέλη. Ε, έγινε, κάποια πρόοδος για αυτό το θέμα και κάποια άλλα, όπως για την προστασία δεδομένων, αλλά δεν επετεύχθη κάποια τελική συμφωνία. Ο επόμενος γύρος του διαλόγου στις 5 Μαΐου 2015, ενώ ε, οι τεχνικές εργασίες εξακολουθούν. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 3. Είναι μεγάλη μας χαρά να υποδεχόμαστε σήμερα τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ε, κύριο Βίτορ Κωνστάνσιο, για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι και η πρώτη φορά που έρχεται ο κύριος Κωνστάνσιο επί νέας θητείας στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και ανεπομονούμε και για τις επόμενες συναντήσεις μας. Η ετήσια έκθεση δημοσιεύτηκε στον επίσημο τοπό της ε, ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μιλάμε για την ε, νομισματική πολιτική και τις οικονομικές εξελίξεις του 2014, καθώς και τις δραστηριότητες του συστήματος του ευρώ στα στους διάφορους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης υπάρχει μια επιστολή που συνοδεύει την έκθεση από τον κύριο Ντράγκη προς τον κύριο Σούλτς με ένα παράρτημα που έχει τις απαντήσεις της ΕΚΤ για τα σχόλια και τι παρατηρήσει τη ε, Έκθεση ιδία πρωτοβουλία 2014 τη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με εισηγητή τον ε, Αντιπρόεδρο κ. Θάλμπα. Η επιστολή αυτή σα έχει μεταβεβαστεί από τη Γραμματεία σήμερα το πρωί. Βάσει του άρθρου 224 τη συνθήκη, συνθήκης, αιτήσια έκθεση τη ΕΚ πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα ετοιμάσει έκθεση ιδέα πρωτοβουλία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 President Draghi, during his last hearing to this committee, already highlighted the efforts οι προσπάθειες που καταβάλει αυτή τη στιγμή η ΕΚΤ για να πετύχει το στόχο της σταθερότητας των τιμών με στόχο πληθωρισμού κοντά στο 2% για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη σωστή ε, υλοποίηση τη νομισματική πολιτική αλλά και την οικονομική ανάκαμψη. Ιδίω η ποσοτική χαλάρωση και σχετική απόφαση της ΕΚΤ και το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού. Πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός μεταβίβασης νομισματικής πολιτική θα προχωρήσει με άλλα τμήματα της εθνική πολιτική, ακόμα και παρά τον χαμηλό ρυθμό της ε, ε, πολιτική το 2014. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει δημοσιονομική σταθεροποίηση ε, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτού του, αυτού πολιτική αυτής της ανάμειξης πολιτικής και την προσπάθεια να υλοποιηθούν οι απαραίτητες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. αλλά και να ε, πετύχει το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αρχίσει να λειτουργεί σύντομα. Θεωρούμε ότι αυτό το περιβάλλον που θα είναι φιλικό προς την ανάπτυξη θα έχει να κάνει και με, την ενώση των αγορών που θα συναντήσουμε σύντομα στην Επιτροπή μας και για τον οποίο θα ετοιμάσουμε και μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Αυτές ήταν οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Επιτρέψτε μου όμως να σας δώσω το λόγο για να περάσουμε και στην ανταλλαγή απόψεων. Ο λόγος τον Αντιπρόεδρο Κωνστανσιο. Και μετά θα έχουμε τις ερωταπαντήσεις. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που είμαι και πάλι σε αυτή την Επιτροπή για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεσή μας. Το, το γεγονό αυτό τονίζει και πάλι τη σημασία του διαλόγου με το Ευρωκοινοβούλιο για να υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια στι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακριβώ, επειδή η ΕΚΤ θεωρεί τη διαφάνεια ένα ζωτικό στοιχείο τη λογοδοσία και τη αποτελεσματικότητα, φέτο αρχίσαμε να δημοσιεύουμε λογαριασμού από τι συνεδριάσεις μα και τι συζητήσει για την νομισματική μα πολιτική. Η δημοσίευση της ετήσιας έκθεση συμπληρώνει τις προσπάθειές μας για μεγαλύτερη διαφάνεια με περιγραφή των δράσεων της ΕΚΤ το 2014 και με σκοπό να εκπληρώσουμε τη θητεία μας σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπως τονίσατε. Η, η δράση της ΕΚΤ ήταν απαραίτητη για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες μεταβίβασης των ε, στοιχείων της νομισματικής μας πολιτικής και το περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού. Και ένα άλλο μεγάλο επίτευγμα το 2014 ήταν οι προετοιμασίες ε, και η έναρξη λειτουργίας του ε, ενιαίου μηχανισμού επιθεώρησης. Εδώ η διαθεσμική συμφωνία μεταξύ ΕΚΤ και Κοινοβουλίου προβλέπει λογοδοσία και για αυτή τη νέα αρμοδιότητα της ΕΚΤ. Σήμερα θα ήθελα να δούμε τα μέτρα που ανέλαβε η ΕΚΤ από την αρχή της περασμένης χρονιάς για να πετύχει τον ε, στόχο της και επίσης ε, θα θέλαμε να συζητήσουμε το, πρόγραμμα, το εγχείρημα της ένεσης κεφαλαίου γιατί εάν υπάρξει απαραίτητη φιλοδοξία θα έχουμε χρηματοπιστωτική ε, ολοκλήρωση και σωστή μετάδοση της νομισματικής μας πολιτικής. Το περιβάλλον της νομισματικής πολιτικής το 2014 ήταν περίπλοκο και απαιτητικό. Η μεταβλητή ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2013 δεν επιταχύνθηκε όπως αρχικά αναμενόταν. Και ολόκληρη τη χρονιά είδαμε το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,9% στην Ευρωζώνη. Η ανάπτυξη αυτή ε, υποφέρει ακόμα, δεν είναι σταθερή και οι πιστώσεις συρρυκνώνονται. Ε, υπάρχει φθήνων ρυθμός και ε, τα πρότυπα για τις πιστώσεις με τα υψηλά επιτόκια της Ευρωζώνης έχουν οδηγήσει σε οικονομική καθυστέρηση στην, σε επίπεδο Ευρωζώνης και είναι ένας λόγος του αποπληθωρισμού για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες της μετάδοσης του μηχανισμού του νομισματικού μας, της νομισματικής μας πολιτικής, εγκρίναμε ένα πακέτο μέτρων τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο. Ε, Επίσης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο υπήρχαν τα εξής τρία βασικά στοιχεία. Ε, οι δύο μειώσεις στα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ με μια τάση να είναι στο χαμηλότερο βαθμό τους και επίσης οκτώ στοχευμένες προσπάθειες μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης καθώς και δύο προγράμματα ε, αγοράς καλυμμένων ομολόγων. Εδώ βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ενδυνάμωσης, όμως ο φθήνων ρυθμός του πληθωρισμού επιταχύνθηκε στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου το δεύτερο εξάμεινο του 2014 ε, ενίσχυσαν αυτήν την ε, εξέλιξη και καταλήξαμε στο τελευταίο μέρος μιας ε, μακροχρόνιας τάσης να είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ο πληθωρισμός με συνέπειες δεύτερο, Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια ε, τάση διατήρησης αυτής της ε, ε, αυτής της πορείας και, το σύστημα του ευρώ, και γι' αυτό το ε, σύστημα του ευρώ αποφάσισε τις 22 Ιανουαρίου του 2015 να προχωρήσει με τα προγράμματα αγοράς και σε αξιογραφά του δημόσιου τομέα. Ε, αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2016 και σε κάθε περίπτωση μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο να δει ότι υπάρχει σταθερή προσαρμογή το κομμάτι του πληθωρισμού και η οποία συνάδει με το στόχο να πετύχουμε ε, ποσοστά πληθωρισμού ε, κάτω ή έστω κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Όλα αυτά, ειδωμένα από κοινού, δείχνουν ότι τα πολιτικά μας μέτρα συμβάλλουν σε χαμηλά επιτόκια στις κεφαλαιαγορές και βοηθούν αυτές οι θετικές εξελίξεις να επικρατήσουν σε όλη την ε, αλυσίδα διαμεσολάβησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις στην μετάδοση των στοιχείων της νομισματικής πολιτικής τη ΕΚΤ στην πραγματική οικονομία. Και αυτό με διευκόλυνση για τι χρηματοπιστωτικέ συνθήκε και τι οικονομικέ συνθήκε των οικοκυριών και των εταιριών και με τη σημαντική πτώση των ε, ε, επιπέδων ε, των επιτοκίων για τα δάνεια και την συρρήκνωση αυτή του κατακαιρματισμού στην Ευρωζώνη. Τα τραπεζικά επιτόκια έχουν πέσει σημαντικά από το καλοκαίρι του 2014 κατά 40 ή για την περίπτωση των οικοκαιριών 50%. Και το ε, ονομαστικό κόστος της εξωτερικής, ε, του εξωτερικού δανεισμού για την Ευρωζώνη έχει μειωθεί περαιτέρω και φτάνει το 4,1% τον Φεβρουάριο. Αυτό θα μπορούσε να προωθήσει και να ενισχύσει την ανανέωση στις πιστώσεις και τις επενδύσεις. Οι πιστώσει των τραπεζών σε μη χρηματοπιστωτικέ εταιρείε αυξήθηκαν του τελευταίου τρει μήνε με ένα ετήσιο επιτόκιο του 2% που θα πρέπει να το συγκρίνουμε με το αρνητικό επιτόκιο της περασμένης χρονιάς που ξεπερνά το μείον 2%. Πράγματι, τον Φεβρουάριο πέρσι ο ρυθμός ε, ανάπτυξης αυτών των πιστώσεων ήταν μείον 0,3% προς τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Καταφέραμε λοιπόν το τελευταίο τρίμενο να έχουμε θετικό πρόσημο στα ποσοστά αυτά εδώ και πολύ καιρό. Ένα γενικότερο κύκλο εργασιών για το τελευταίο τρίμηνο του 2014 για τι μη χρηματοπιστωτικέ εταιρείε ήταν ε, μια σημαντική αύξηση. Επίση, η ε, ε, σταθερή αύξηση του M1 οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη κατά την προοπτική αυτή. Αυτή η αξιολόγηση, όπως δείχνει η σχετική έρευνα για την Ευρωζώνη, ενισχύει τις δυνατότητες ε, δανειληψίας για τα νοικοκυριά και τις εταιρείε και βελτιώνει τις ε, προϋποθέσεις ε, χορήγησης πιστώσεων. Αυτές οι πολιτικές με την οικονομική μας ανάπτυξη φαίνεται να γίνονται ε, αρκετά αυτοματοποιημένες και το αρνητικό, ε, η αρνητική αυτή απόσταση μάλλον θα καλυφθεί μέχρι το 2017. Έτσι, οι προσδοκίες μας περί πληθωρισμού φαίνεται ότι θα συνάδουν τελικά με την εντολή που λάβαμε παρά το ε, τράνταγμα της αλλαγής της τιμής του πετρελαίου και την προσπάθεια να ε, εξομαλύνουμε τον πληθωρισμό στα πρώτα στάδια. Αλλά ε, η νομισματική μα πολιτική δεν λειτουργεί μόνη τη. Υπάρχουν και άλλε πολιτικέ πρωτοβουλίε που είναι εξίσου σημαντικέ. Γι' αυτό το λόγο η έναρξη λειτουργία του ενιαίου μηχανισμού επιθεώρηση και ε, η ολοκλήρωση της ε, συνολικής ε, αποτίμησης ήταν καθοριστικά βήματα για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια υγιέστερη νομισματική πολιτική και την ε, σωστή της μετάδοση. Γενικώ, ο μηχανισμός επιθεώρησης και η Τραπεζική Ένωση σε συνδυασμό με τις δράσεις του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης και του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης είναι στοιχεία που θα συνεισφέρουν περαιτέρω στην κατάργηση του φαύλου κύκλου μεταξύ του κρατικού χρέου και των αναγκών των τραπεζών. Χρειάζεται εδώ μια σφαιρική στρατηγική όμω για να δημιουργήσουμε τι προποθέσει για μια σταθερή ανάκαμψη που να βασίζεται στι επενδύσει, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση και την ανάπτυξη τη πραγματικότητα. Οι δημοσιονομικέ πολιτικέ θα πρέπει να στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη και να διασφαλίζουν την βιωσιμότητα του χρέου. Ταυτόχρονα οι διευθυντικέ μεταρρυθμίσει θα πρέπει να υλοποιούνται ε, εγκαίρω και με πυγμή, οπότε οι εταιρείε και τα νοικοκυριά να είναι όχι απλώ σε θέση, αλλά και πρόθυμα να επενδύσουν. Θα πρέπει να επαναλάβουμε αυτή την έκκληση, διότι ο συνδυασμό τη σωστή δημοσιονομική πολιτική και των βελτιωμένων οικονομικών ε, δομών μπορεί να κάνει την νομισματική πολιτική πιο αποτελεσματική και να ενθαρρύνει του οικονομικού φορεί να ε, αξιοποιήσουν τις βελτιωμένες ε, συνθήκες της οικονομίας και να επενδύσουν περισσότερο. Η νομισματική πολιτική μπορεί και θα εξομαλύνει και επιταχύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και δεν μπορεί βεβαίως, ε, αλλά δεν μπορεί βεβαίως να απογειώσει αυτή την προσπάθεια. Έτσι χρειάζονται και πόροι οι οποίοι να προβλεφθούν και να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά. Προ αυτό το στόχο η Ένωση Κεφαλαιογορών και το σχετικό πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει σοβαρά στην όλη προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σκοπεύει να προβλέψει τα βασικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιογορών στην διάρκεια της ε, τρέχουσας θητεία. Από τη δική μα την προοπτική ένα τέτοιο εγχείρημα εφόσον είναι ε, συνολικό και σωστά σχεδιασμένο μπορεί να φέρει σοβαρά ωφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση Κεφαλαιογορών είναι ένα μέσο για να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση των κεφαλαίων αγορών, βεβαιωνόμενοι ότι αυτή η ολοκλήρωση θα γίνει εύρωστη. Οι ε, ε, ενωμένε κεφαλαίων αγορέ μπορούν να ενισχύσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα ε, με την κατανομή του ιδιωτικού κινδύνου και να βελτιώσουν την απορρόφηση των κραδασμών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, οι εύρυθμε κεφαλαίε μπορούν να βελτιώσουν και τη μετάδοση τη νομασματική μα πολιτική. Η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση είναι κάτι που ούτω ή άλλω αναφέρεται και στο, στη δήλωση για την εντολή του ευρωσυστήματο. Η Ένωση Κεφαλαίου είναι ένα πρόγραμμα για την διαφοροποίηση και το μέγεθο των κεφαλαίων αγορών με περαιτέρω εξέλιξη συγκεκριμένων τμήματων τη αγορά η βαθύτερη και περισσότερο διαφοροποιημένη αγορά κεφαλαίων μπορεί να προβλέψει και περισσότερε πηγέ χρηματοδότηση όπω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τα έργα υποδομών ή την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα η μείωση τη οικονομική εξάρτηση από την χρηματοδότηση των τραπεζών μπορεί να μα προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων για την σωστή διεξαγωγή τη νομισματική μα πολιτική. Ωστόσο, υπάρχει ένα πραγματικό κίνδυνο να υπάρξει αποτυχία να εντοπίσουμε τι σωστέ προποθέσει ώστε να πετύχει του στόχου τη Ένωση των Κεφαλαίων Α είμαστε σαφεί. Ε, μια πραγματική ένωση κεφαλαίου αγορών σημαίνει ένα υψηλό επίπεδο χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και την ε, ε, εδραίωση τη ενιαία αγορά σε αυτόν τον τομέα. Σε μια πραγματική ένωση κεφαλαίου όλοι οι φορεί τη αγορά θα πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ε, για να ε, είναι αντιμέτωποι με ένα ε, παρόμοιο σύνολο κανόνων. Να έχουν την ίδια πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τι υπηρεσίε και να την χάνουν ίδια μεταχείριση όταν δρουν στην αγορά. Η Ένωση Κεφαλαίου της τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κοινό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που, προσφέρει, ε, που προβλέπει μάλλον ίδιους κανόνες και επιτρέπει στις αγορές να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν. Αυτό βεβαίως έχει μια σειρά από επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα ο στόχος του να έχουμε μια ένωση κεφαλαίου αγορών είναι από μόνος του πολύ φιλόδοξος. Ελπίζουμε ότι αυτή η ένωση θα πετύχει τα ε, αποτελέσματα που θέλουμε χωρίς να υπάρξει όμως πλήρη ε, πλήρης εναρμόνιση, κάτι που θα ήταν απλώς ευσεβής πόθος. Το να καταφέρουμε τα περισσότερα από τους στόχους μας είναι ήδη αρκετό. Ε, το να υπάρξει πλήρης ε, ένωση κεφαλαίου αγορών δεν είναι ένωση κεφαλαίου αν το πετύχουμε κατά το ίμιση. Αυτό φαίνεται και από τα διδάγματα της κρίσης, διότι υπάρχει ε, αλληλεπίδραση μεταξύ της ενίας αγοράς και του πλημελούς ρυθμιστικού και εποπτικού ε, πλαισίου. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα για τις ε, κεφαλαίες αγορές. Επίσης το να υπέρχει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τις κεφαλαίες αγορές και όλους τους τομείς της πολιτικής που μας ενδιαφέρουν με τους φραγμούς που μπορεί να προβλέπουν είναι κάτι που θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια των κεφαλαίων αγορών. Αυτό αφορά πολιτικά ευαίσθητους τομείς όπως την αφαιρεγγιότητα ή τους νόμους για το επιχειρηματικό κεφάλαιο, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί τώρα νομοθετική πρόοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειαστεί τουλάχιστον συντονισμένη δράση σε εθνικό επίπεδο για να περιοριστούν οι κρατικοί φραγμοί. Επιπλέον, το ενιαίο σύνολο κανόνων θα πρέπει να συμπληρωθεί ε, εν καιρό από κοινή υλοποίηση και επιβολή των κανόνων γιατί υπάρχει μεγαλύτερος αλληλοσυσχετισμός ε, από την Ένωση Κεφαλαίου Αγοράν αγορών που θα αυξήσει τους κινδύνους ε, ε, μόλυνσης των στοιχείων αυτών της αγοράς και θα επηρεάσει την εποπτεία των αγορών από τους σχετικούς φορείς. Το Ευρωκοινοβούλιο ως σύνομοθέτης έχει ένα καθοριστικό ρόλο διαδραματίσει εδώ σε αυτή τη διαδικασία και ελπίζω ότι θα συνεισφέρεται τα μάλα στη δημιουργία μιας πραγματικής ένωσης κεφαλαίου αγορών. Να ολοκληρώσω. Ε, οι βασικέ προσπάθειε που έχουν αναλυθεί από την αρχή του 2014 σε ό,τι αφορά και την νομισματική πολιτική και την ε, τραπεζική ένωση δείχνουν ότι η Ευρώπη ε, μπορεί να πετύχει αποτελέσματα όταν χρειάζεται αποφασιστική δράση. Ωστόσο πρέπει να πάμε παραπέρα η εύρωστη δημοσιονομική και διαθωτική πολιτική σε εθνικό επίπεδο είναι τα περαιτέρω βήματα για να ενισχύσουμε τη θεσμική ε, σωστή παρακολούθηση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να μπορέσει η οικονομία τη Ευρωζώνη να γίνει πιο αντακτική. Επίση, οι αποφασιστικέ δράσει και μεταρρυθμίσει χρειάζονται για να στηρίξουμε τη δημιουργία μια πραγματική Ένωση Κεφαλαίου Αγορών με σκοπό να απελευθερώσουμε όλο το δυναμικό αυτή τη ευρωστότερη ε, οικονομική ολοκλήρωση. Αυτέ οι εξελίξει θα χαράξουν το δρόμο για μια σταθερή ανάκαμψη και μια ισχυρότερη νομισματική ένωση που να είναι ανθεκτικότερη στους ε, κραβασμούς και να εγγυηθεί την σταθερότητα και την ευημερία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε Κωνσταντσιο. Πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ήταν πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών που τα χρειαζόμαστε γιατί αυτό συζητούμε και συμφωνούμε απόλυτα ότι αν θέλουμε πραγματικά μια Ένωση Κεφαλαίου Αγορών και τα ωφέλη της θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη την ανάγκη της ε, πλήρους κανονιστικής εναρμόνισης. Πολύ χρήσιμη αυτή η παρατήρηση. Και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη γιατί πρέπει να διαβάσω την Προεδρία στον Πίτερ Σάιμον γιατί πρέπει να ετοιμαστώ για την ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ακολουθήσουμε λοιπόν ε, την ε, συνηθισμένη διαδικασία. Πέντε λεπτά για ερωτοπαντήσει. Καταρχά για όλε τι ομάδε και για του μη εγγεγραμμένου και στη συνέχεια με το σύστημα DONT. Με το ΕΛΚ e θα ξεκινήσουμε. Ο κύριο Σουμποκατμπάλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κωνσταντσιο. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα θίξατε σήμερα. Θα μπορούσαμε πολλά να επιλέξουμε να θίξουμε. Εγώ τρει ερωτήσει έχω, αρκετά σύντομε, να σα θέσω. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την επιτοκή πολιτική του ΕΚΤ, οι πάροχοι μακροπρόθεσμων προϊόντων όπως ε, οι ασφαλίσεις βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν φοβάται η ΕΚΤ εδώ να δημιουργήσει μια νέα κρίση περιουσιακών στοιχείων παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα περάσει την τραπεζική κρίση. Δεύτερη ερώτηση. Η εξάντληση της αγοράς ομολόγων με τις διαρκές αγορές της ε, ΕΚΤ. Αυτό ενισχύει τις ε, τη, τις ε, διαφορές στην τιμή, στις τιμές. Πώς θέλετε λοιπόν να αποτρέψετε αυτές τις τάσεις. Και τρίτη ερώτηση σε ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις των τιμών. Τρίτο θέμα. Η ρευστότητα. Σίγουρα αποτελεί ένα θέμα για, την αρνητική, για τα αρνητικά ε, επιτόκια στους πιστωτές. Πιστεύετε ότι αυτά είναι επιθυμητές διαδικασίες ή μήπως αυτό καταδεικνύει ότι έχουμε περβεί κάποια διασυνοριακά εμπόδια σε ό,τι αφορά αυτές τις συναλλαγές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Να ξεκινήσω απαντώντας και σχολιάζοντας το εξής, όλες οι πολιτικές έχουν ε, αρνητικά και θετικά και κάποιες δευτερευτούσες συνέπειες, κάποιες απευκτές αλλά δυστυχώς και αναπόφευκτες αν οι προτεραιότητες μας οδηγούν να κάνουμε κάποιες επιλογές στις πολιτικές μας. Αυτό ακριβώς λοιπόν συμβαίνει και συνέβη και το περσινό έτος ε, ο πληθωρισμός ε, πήρε αρνητικό πρόσημο και να σημειώσω ότι στο δεύτερο ήμιση του έτους ο πληθωρισμός επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη μείωση των πετρελαϊκών τιμών, αλλά το Δεκέμβριο και τώρα αναγνωρίζουμε το πόσο συνέβαλε η τιμή του πετρελαίου στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι 0,6, στο 0,6. Απέχει πολύ λοιπόν και βασίζεται στις εγχώριες πραγματικότητες. Απέχει λοιπόν πάρα πολύ από την εντολή μας και από το στόχο μας. Άρα έπρεπε να λάβουμε μέτρα έπρεπε να λάβουμε μέτρα τα οποία φυσικά είχαν επεκτατική φύση, προσπαθώντας να καλύψουν το κενό της παραγωγής στην, ε, στην ζώνη ευρώ και να μειώσει τις προσδοκίες που, να αντισταθμίσει τις προσδοκίες που έπεφταν. Αντιλαμβανόμαστε τις ενδεχόμενες συνέπειες μιας πολιτικής τέτοια στις ε, αγορές ε, στοιχείων, αλλά δεν είχαμε επιλογή και αναπτύσσουμε μία ανάλυση του τι συμβαίνει, παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά. Είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε μακροοικονομικά μέτρα για να περιορίσουμε τον κίνδυνο στις αγορές αυτές ε, στοιχείων σε ό,τι αφορά τις ε, ασφάλειες. Να επισημάνω το εξή. Τα τελευταία τρία χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια, η απόδοση στις ε, ασφαλιστικές ήταν στο 9%, πολύ πιο υψηλό ποσοστό από τις τράπεζες. Τα τελευταία τρία χρόνια η έσοδα αναμετοχή των ασφαλιστικών ήταν πολύ υψηλότερα και πάλι από ό,τι οι τράπεζες. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Για δύο λόγους βασικά. Καταρχάς, οι ασφαλιστικές ε, εποφελούνται από τα κέρδη των κεφαλαίων όταν μειώθηκαν οι αποδόσεις και από τις τιμές ε, των στοιχείων που ανέβηκαν. Το, κατά δεύτερον, το γεγονός ότι είναι τόσο χαμηλός ο πληθωρισμός επηρεάζει και τον υπολογισμό των ευθυνών των ασφαλιστικών. Άρα, ανησυχούμε, δεν λέω, ότι μακροπρόθεσμα, αν τα κέρδη αυτά, τα κεφαλαιακά, μειωθούν, μπορεί να δημιουργηθεί πίεση από τα επιτόκια, αλλά δεν έχουμε ακόμα φτάσει στην κατάσταση αυτή. Αυτό λοιπόν ήθελα να θα τονίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις ε, και σε πόσο επηρεάζουν οι πωλήσει στις τιμές. Είμαστε προσεκτικοί για να μειώσουμε και να περιορίσουμε τις αγορές μέσα στο 33% κατά το όριο σε ό,τι αφορά το χρέος του κάθε ασφαλισμένου. Αυτό τι σημαίνει ότι ε, επιτρέπουμε και ένα περιθώριο να λειτουργήσει και η αγορά. Να επηρεάσει την ελεύθερο καθορισμό τιμών στην αγορά. Δεν είμαστε οι μόνοι φορείς στην αγορά σε καμία περίπτωση. Το γεγονός ότι κάποια επιτόκια κινούνται σε αρνητικά πρόσημα είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε στόχο μας. Θέλαμε να μειώθουν τα επιτόκια και άλλο, αλλά όχι απαραίτητα να κινηθούν με αρνητικά πρόσημα. Είναι δευτερεύουσα συνέπεια και αυτό γύρει και ερωτήματα για το πώς διαμορφώνονται οι προσδοκίες ε, της αγοράς σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Τα βραχυπρόθεσμα λοιπόν επιτόκια να κινούνται σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Αυτό όμως και πάλι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν θα συνεχιστεί στους ίδιους ρυθμούς. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ελπίζουμε σύντομα να το διορθώσει η αγορά αυτό. Σας ευχαριστώ. Η Ελίζα Φαρέιρα για το επόμενο χρόνο διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που Πολλές φορές αγκομίασα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη γνώμη του θεσμικού όργανο που έδειξε τη μεγαλύτερη ικανότητα στην αντιμετώπιση της κρίσης. Έχω τώρα δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά αυτό που μας είπατε και εσείς, το ρόλο της Ένωσης Κεφαλαγορών ως σταθεροποιητικού στοιχείου. Τρία επίπεδα έχουμε εδώ. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Και είναι φυσικό να γίνονται κάποιε προσαρμογέ και κάποιε διορθώσει. Αρχίζουμε όμω και αντιλαμβανόμαστε ότι ίσω ο αντίκτυπο στι ε, περιφερειακέ χώρε για κεφαλαϊκέ απαιτήσει προκαλεί υπερβολική τραπεζική συγκέντρωση που δεν ήταν αρχικά στόχος αυτής της διαδικασίας και γιατί καθιστά το σύστημα πιο τρωτό, πιο ευάλωτο. Σε ό,τι αφορά ε, το θέμα της εξυγίασης, ε, υπάρχει δυνατότητα ενός μηχανισμού αναστολής, ενός ε, backstop και υπάρχει δυνατότητα από τον Ιανουάριο του χρόνου να εξασφαλιστεί η, σταθερο, η σταθερότητα ε, του τραπεζικού συστήματος σε μια διαδικασία εξυγίασης. Και ένα τρίτο στοιχείο, η κοινή εγγύηση καταθέσεων. Έχει εξαφανιστεί αυτό από το πακέτο, παρόλο που είναι ουσιαστικό στοιχείο σταθεροποίησης της αγοράς και αποτελούσε τμήμα του αρχικού πακέτου. Είναι θέμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Δεν μπορεί να εξαφανίζεται έτσι με μια μονοκοντιλιά από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ε, παρέσει ήταν σιωπηλό ε, και διακριτικό προ το θέμα αυτό. Γιατί επίση ε, υπάρχει μια μακροοικονομική ανισορροπία αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σε πια τιμέ δεν έχουν αξία οι, μέσες, ε, οι μέσοι δείκτες. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο γιατί έχουμε μια Ευρώπη με υψηλά επίπεδα ανεργία και στασιμότητα. αλλά αυτά τα φαινόμενα πλήττουν περισσότερο την μισή Ευρώπη. Στην υπόλοιπη δεν γίνονται αισθητά. Έχει επίγνωση αυτή τη μακροοικονομική ανισορροπία ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πώ πιστεύετε ότι το ελληνικό πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει την Ευρωζώνη, γιατί είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στα αγγλικά γιατί θα είναι πιο εύκολο για τους υπόλοιπους ε, να με καταλάβουν. Καταλαβαίνω ότι εσείς τη μητρική σας ε, που είναι και δική μου, τα πρωτογαλλικά, αλλά λόγω συνήθειας για μένα είναι ευκολότερο για τα τεχνικά θέματα να χρησιμοποιώ την αγγλική γλώσσα και όχι τη μητρική μου. Και σας ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα συνεχίσω στα αγγλικά. Πάντως έχετε δίκιο ότι είναι πολύ σημαντική η Τραπεζική Ένωση και αυτό που είπατε, ο κίνδυνος συγκέντρωσης ε, των τραπεζικών. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, δεν έχουμε τέτοια παράδειγμα διασυνοριακών αγορών ή διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Πάντως, ε, πολύ πιθανόν να συμβούν κάποιες τέτοιες, να συμβούν κάποιες τέτοιες συγκεντρώσεις. Ήταν αφέλες να το αγνοούμε. Γιατί υπάρχουν κάποια σημεία ε, στην Ευρώπη που η κατάσταση δικαιολογεί μια τέτοια συγκέντρωση. Ιδιαίτερα μια στιγμή που βλέπω μια μετάβαση ε, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τις ε, τραπεζικές δραστηριότητες σε χρηματοδότηση που στηρίζεται στις αγορές. Αυτό συμβαίνει και φυσικά δημιουργεί νέους κινδύνους αλλά και νέο ωφέλη γιατί διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεταστροφή κατά κάποιο τρόπο και καλό θα ήταν να έχουμε κάποια εδραίωση στην πορεία. Σε ό,τι αφορά το backstop και την εξυγίαση, resolution, φυσικά έχουμε έναν εκπρόσωπο με θέση παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μηχανισμού Εξυγίασης και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τα θέματα και αν όντως η κατάσταση ε, καταστήσει απαραίτητη αυτή την προϋπόθεση θα επιμείνουμε στη συμφωνία ότι ο μηχανισμός και η αρμόδια αρχή για την ε, εξυγίαση των τραπεζών θα πρέπει να έχει και αυτή την ε, γραμμή τη χρηματοδότηση. Ό,τι αφορά το σύστημα εγγύηση καταθέσεων, αυτό το αναφέραμε ανέκαθεν ως το τρίτο στοιχείο της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Βέβαια δεν είχαμε ευκαιρία να το αναλύσουμε, αλλά επιμείναμε και η επιλογή των κρατών μελών ήταν να αναβληθεί η εφαρμογή αυτή, αυτού του τρίτου άξονα της Τραπεζικής Ένωσης. Οπότε διαπιστώνουμε ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο για το θέμα αυτό, για αυτό, το, για αυτό το θεμέλιο, αλλά σίγουρα δεν το έχουμε ξεχάσει το θέμα του ε, κοινού συστήματο εγγύηση καταθέσεων. Σε ό,τι αφορά του μέσου όρου και τι ανισορροπίε, έχετε απόλυτο δίκιο, ιδιαίτερα για την ανεργία. Στα θέματα ανεργία, οι διαφορέ μεταξύ των χωρών μελών είναι τεράστιε. Αλλά η κατακαιρμάτιση όλους τους έχει, ο κατακαιρματισμό σε όλους του άλλου τομεί έχει μειωθεί και σε θέματα ανάπτυξης γιατί έχουμε κάποιες χώρες περιφέρειας που αναπτύσσονται με ρυθμούς ψηλότερους από τους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης. Κάτι που σημαίνει ότι ο κατακαιρματισμός, ακόμη και από αυτή την άποψη, της ε, οικονομικής μεγέθης κάπως διορθώνεται. Οπότε υπάρχει μια βελτίωση και θα έλεγα ότι οι πολιτικές μας συνέβαλαν σε αυτή τη μείωση του κατακαιρματισμού στην Ευρώπη. Um- σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δώσουμε σε όλου του αδέλφους την ευκαιρία να μιλήσουν, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να περιοριστούμε στο χρονικό περιθώριο 5 λεπτών. του Λούκε από το ECR τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για την προθυμία σα να απαντήσετε στι ερωτήσει. Θα ήθελα να συνεχίσω την ερώτηση τη Γερίζα Φεραίρα για την ε, κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν είναι σαφέ κατά πόσον η Ελλάδα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πληρωμών τη τον Μάιο. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές και πάλι. Πώς ε, αξιολογεί η ΕΚ την κατάσταση αυτή και θα μπορούσατε ενδεχομένως ε, να δώσετε μια υπόσχεση ότι η Ελλάδα δεν θα καθεστεί αφρέγγια λέγοντας ότι για παράδειγμα θα υπάρξει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αν δεν μπορείτε να δώσετε, για την Πρόεδρε, μια τέτοια υπόσχεση, θα ήθελα να μου πείτε, επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια και για την εποπτεία, την τραπεζική, κατά πόσον συμβουλεύετε τις ε, ελληνικές ε, τράπεζες να αποχωριστούν τα ευρωπαϊκά ομόλογα, να αφήσουν τα T-bills, προκειμένου σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας του ελληνικού κράτους να είναι μικρότερη η επίπτωση της ελληνικής τράπεζας. Και κατά τρίτον, θα θέλω να μας πείτε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει οποιαδήποτε σχέδια και προγραμματισμό για ένα ενδεχόμενο, ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ. Υπάρχει λοιπόν κάποια προετοιμασία για την περίπτωση που η Ελλάδα δεν θα παραμείνει, δεν θα μπορέσει να παραμείνει στο ευρώ, στην ευρωζώνη αν ε, καταστεί αφαιρέγγια η Ελλάδα ή πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται μια τέτοια προετοιμασία γιατί μια ελληνική αφαιρεγγιότητα του κράτους, δηλαδή της Ελλάδας, δεν θα θέσει ένα αμφιβόλο την συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Μπορεί δηλαδή να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη ακόμα και αν ε, δεν είναι, είναι αφαιρέγγια η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας αυτές για ένα πολύ σημαντικό τέτοιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν πάντα ανοιχτή σε ό,τι αφορά την επικοινωνία των κανόνων της για τη χρηματοδότηση του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, στην παρούσα φάση το σύνολο, το συνολικό ποσό ρευστότητας, το οποίο έχει χορηγηθεί από το σύστημα της Ευρωζώνης, από το, στις ελληνικές τραπέζες, ανέρχεται στα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι περίπου στο 70% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Είναι λοιπόν δύσκολο να πούμε ότι δεν έχουμε χρηματοδοτήσει τις ελληνικές τράπεζες. Γιατί η ΕΚΤ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το τμήμα του SSM της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες είναι φερέγγιες. Αυτό λοιπόν είναι πρώτη υπόθεση για να δοθεί πίστοση. Δεν ήταν αυτή η ερώτηση, λέει ο κύριος Μπέντ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Συμπεραίνω λοιπόν το εξή. Ότι ήμασταν πάντα ανοιχτοί, δεν μπορώ όμως να σας υποσχεθώ, όπως το γνωρίζετε και το φαντάζεστε, και αυτό το υπονοεί και η ερώτησή σα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα χρηματοδοτήσουμε την Ελλάδα οτιδήποτε και αν συμβεί, οποιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση, ανεξαρτήτω όρων. Υπάρχουν κανόνε. Ένα από του κανόνε σχετίζεται με την, το να υπάρχουν εγγυήσει στι τράπεζε, ασφάλειε στι τράπεζε. Ε, Αναφέρατε στην ε, απάλυνση ή στην κατάργηση ενδεχομένως ε, της σχέσης μεταξύ τραπεζών και, τραπεζών και κράτους. το SSM έχει προτείνει και το Αντικτικό Συμβούλιο της ε, ΕΚΤ έχει εγκρίνει οι ελληνικές τράπεζες να μην αυξήσουν από εδώ και πέρα την έκθεσή τους στο ελληνικό κράτος. Να μειώσουν. Αυτό δεν αποφασίστηκε. Αποφασίστηκε να μην αυξηθεί η έκθεση. Περαιτέρω. Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθησε που προστατεύει την φρεγγιότητα των τραπεζών στην τρέχουσα φάση με επιτόκια και κεφαλαιοικά που είναι σημαντικά θετικά. Και αυτό λοιπόν έχει συμβεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χειρότερο σενάριο, δεν θέλω να κάνω εικασίες, γιατί είμαι πεπισμένος και είμαστε πεπισμένοι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν θα υπάρξει έξοδος της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο δηλαδή που θα φέρει την Ελλάδα εκτός ευρώ. Όπως ξέρετε, η συνθήκη δεν προβλέπει μια χώρα να αποχωρήσει νόμιμα, να διωχθεί νόμιμα από το ευρώ. Άρα, σε τελική ανάλυση, μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση και όχι από εμάς δεν είναι μία εικασία τέτοια. Δεν υπάρχει εικασία ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Και θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί. Δεν είναι δε αυτόματο ότι μία εγκαιότητα του ελληνικού κράτους προς ένα πιστωτή δεν σημαίνει αυτό αυτόματα ότι η Ελλάδα θα βρεθεί εκτός ευρώ. Από την Άλτε τώρα η Σιλβιγκουλάρ. Καλημέρα σας κύριε Αντιπρόεδρε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Εγώ δεν θα σας θέσω ερωτήσεις για την Ελλάδα, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορείτε και να απαντήσετε. Ας είμαστε πιο επικοδομητικοί όμως. Σας ανησυχεί η μείωση των επιτοκίων και κυρίως ο αντίκτυπος αυτής της μείωσης στον τομέα των ασφαλιών, ασφαλιών ζωής. Και συμπληρωματική ερώτηση στην αναγγελθήσα Ένωση Κεφαλαιογορών δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το φορολογικό σκέλος, γιατί είναι εμφανές ότι η αποταμίευση που είναι πληθωρική στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ε, περισσότερο προσανατολίζεται ε, σε αγορά ομολόγων. Προσανατολίζεται παρά σε αγορά μετοχών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες, Ήδη έχω απαντήσει ένα τμήμα της ερώτησης προηγουμένως. Είπα ότι η κατάσταση και τώρα και στο πρόσφατο παρελθόν, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο για τις τράπεζες. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για τις ασφάλειες από ό,τι για τις τράπεζες. Τώρα, για το άλλο θέμα, ναι, αν δεν αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον, ένα περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια ίσως δημιούργησε περαιτέρω πιέσεις της ασφάλειας και ιδιαίτερα της ασφάλειες ζωής όπως είπατε κι εσείς. Αυτό όντως ισχύει. Και περιμένουμε, και αυτό δείχνουν και προσωμιώσεις που κάνουμε, ότι από το 2017 ε, η κατάσταση θα αλλάξει. Και σίγουρα αν ο πληθωρισμός φτάσει γύρω στο 2% και τα επιτόκια θα αρχίσουν να αυξάνονται. Οπότε θα αλλάξει αυτό το περιβάλλον των ε, χαμηλών, πολύ χαμηλών επιτοκίων. Γιατί στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε αυτό το 2% του πληθωρισμού. Αυτό είναι το επιθυμητό. Επίσης, εδώ έχουμε ένα περιβάλλον που σχεδόν είναι γενικευμένο. Παγκοσμίω ισχύουν χαμηλά επιτόκια, που σημαίνει ότι και οι προηγμένε οικονομίε για μεγάλο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσουν αυτό το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων. Οπότε οι ασφαλιστέ και άλλα ιδρύματα θα πρέπει τι ευθύνε του, τι υποσχέσει του, τι υποχρεώσει του, τα στοιχεία του παθητικού του να τα ευθυγραμμίσουν με το περιβάλλον αυτό. Και οι υπόπτες θα πρέπει να επεμβαίνουν και να φροντίζουν να μην, να μην υπόσχονται 6% αποδόσεις οι εταιρείε. Θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να αποφεύγονται τις καταστάσεις οι επόπτες. Είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα τις ίδιες εταιρείε και τους επόπτες που θα μεριμνούν. Σας ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ η Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντσιο για την προσέλευσή σας. Είμαι από εδώ. Είναι μια πρώτη συζήτηση αυτή για την έκθεση, την ετήσια έκθεση των δράσεων της ΕΚΤ για το 2014 και διερωτώ με το πρόγραμμα προσαρμογής για την Πορτογαλία, πού ε, καλύπτεται. Διότι το 2014 ήταν ε, ακόμα η Τρόικα στην Πορτογαλία. Και στην έκθεση αυτή δεν φαίνεται να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Είχαμε 78 δις ευρώ δάνειο προς την Πορτογαλία. Και στο κομμάτι του 2014 δεν βλέπουμε καμία αξιολόγηση για το σχετικό πρόγραμμα. Και είναι πολύ περίεργο αυτό γιατί υπάρχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες στην ίδια έκθεση για άλλα θέματα, όπως ε, την αλλαγή έδρας της ΕΚΤ. Με δημοσιονομική επιβάρυνση να τονίσω εν παρόδο. Όμως μιλάμε για ένα πρόγραμμα που είχε σοβαρές επιπτώσεις στην Πορτογαλία, όπως μείωση 5% του ΑΕΠ. Οι 300.000 θέσεις εργασίας που καταστράφηκαν. με 29% ε, ε, το δημόσιο χρέος ε, πιο ψηλά από ό,τι προβλεπόταν. Εδώ λοιπόν δεν βλέπουμε καμία τέτοια λεπτομέρεια, ενώ έχουμε αλλού για άλλα θέματα λεπτομερέστατες πληροφορίες. Ε, το αναγνωρίζετε το θέμα αυτό ως έλλειψη. Και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε μια αξιολόγηση της, έκτης στην, της έκθεση δρασεών σας για όσα έγιναν στην Πορτογαλία. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Να ξεκινήσω θυμίζοντας σε όλους ότι από τα 78 δις που δόθηκαν στην Πορτογαλία, εμείς δεν δανείσαμε ούτε ένα ευρώ. Διότι δεν συμμετείχαμε στην ε, δανεικότητα των κυβερνήσεων. Τα κονδύλια αυτά διατέθηκαν στην Πορτογαλία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα κρατή μέλη, από εμάς. συνεργαζόμαστε με την Τρόικα, τέλος πάντων όπω θέλετε να ονομάσετε αυτόν τον διακανονισμό, σε συνεργασία ε, με την Επιτροπή ε, από νομική σκοπιά. ο Ευρωπαϊκός, το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο που είναι υπεύθυνο για αυτά τα προγράμματα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εκείνη υποπτεύει την υλοποίησή τους. Αυτός είναι ο λόγο που δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία στο φιλοσυλλογισμό. Γιατί δεν δανείσαμε χρήματα στην Πορτογαλία σε καμία άλλη χώρα ούτως ή άλλως. Ε, στο πλαίσιο τέτοιων προγραμμάτων. Επίση, όπως είδατε, η ετήσια έκθεση φέτος και περασμένες χρονιές δεν αναφέρεται την συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την πρόοδο διαφόρων χωρών. Ουδέποτε έχει περιληφθεί, ουδέποτε θα, ε, θα συμπεριληφθεί ούτως ή άλλως. Θα ήταν δηλαδή κάτι το νέο να περιληφθεί σε αυτή την έκθεση. Όταν βεβαίω συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, ερχόμαστε για να εξηγήσουμε τι κάναμε και πώ συμμετείχαμε σε μια συνολική προσπάθεια, αλλά δεν είναι η έκθεση αυτή το σημείο που θα αναλύσουμε αυτέ τι δραστηριότητε. Αυτοί είναι και οι λόγοι για του οποίου δεν βρίσκεται λεπτομέρειε όσων αναφέρατε στην έκθεσή μα. Σε ό,τι αφορά την παρόδο παρατήρησή σα για το νέο κτίριο, τι νέε μα εγκαταστάσει, να θυμίσω ότι υπάρχει μια γενική σύσταση από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο προς όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που θα πρέπει να έχουν δικό τους κτίριο αντί να ε, μισθώνουν ή να νοικιάζουν. Διότι μακροπρόθεσμα κοστίζει λιγότερο από το να πληρώνουμε νίκια. Αυτή ήταν η σύσταση που απλώς ακολουθήθηκε και γι' αυτό το όλο εγχείρημα ολοκληρώθηκε. Δεν ήταν κάτι που αποφασίσαμε εν εθρία ή απομονώ. Συγχωρείτε. 10 δευτερόλεπτα αν γίνεται. Στην ετήσια έκθεση δεν γίνεται η απο μονο συγχωρειτε δεκα δευτερολεπτα αν γινεται στην ετησια εκθεση δεν γινεται η αξιολογηση των αρμοδιοτήτων τη ΕΚΤ στα πλαίσια τη Τρόικα. Ε, πού θα γίνει η αξιολόγηση. Διότι με συγχωρείτε, αλλά θα διαφωνήσω. Η αξιολόγηση των προσαρμογών των χωρών γίνεται σε όλε τι ετήσιε εκθέσει. Με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω τίποτα να συμπληρώσω. Η έκθεση έχει ελεγχθεί είναι και λίγο ε, συντομότερη από τις περασμένες χρονιές. Δεν υπάρχει καμία μνήμα για την Πορτογαλία ή για καμιά άλλη χώρα, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Κύπρο, ούτε καμία άλλη. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Δεν είναι αυτό το σημείο που θα λυθεί αυτό το θέμα. Ούτε θα γίνει αυτή η ανάλυση, ούτε και αυτή η συζήτηση. Ε, Επόμενος, ε, το λόγο στον να σας παρακαλέσω μάλλον να τηρήσουμε το χρονικό όριο των 5 λεπτών και θα ήθελα να σας πω ήδη τώρα ότι αν έχουν, ε, όταν ακούσουμε όλες ε, τις ομάδες και τους μη εγγεγραμμένες θα περιοριστούμε στα τρία λεπτά. Γιατί έχουμε και ψηφοφορίες και μετά τις ε, ψηφοφορίες έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχων Προϋπολογισμού. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο. Έρνες Ούρτασον. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Κωνστάνσιο. Ένα από τα σενάρια που αντιμετώπισε η τράπεζα τα τελευταία χρόνια είναι η πιθανή στάση πληρωμών εκ μέρους μιας χώρας μέλους. Ερωτώ λοιπόν, σε περίπτωση που μια χώρα σταματήσει να πληρώνει, να πληρώνει τις υποχρεώσεις, θα συνεχίσετε τη ρευστότητα γιατί αν έχουμε μια τράπεζα που πλήρει τις προϋποθέσεις, κεφαλαϊκές απαιτήσει, όλες τις προϋποθέσεις που βάζεται σε μια εμπορική τράπεζα, σε περίπτωση στάσης πληρωμών της χώρας θα συνεχίσετε να χορηγείτε ρευστότητα σε, αυτό το, σε αυτές τις τράπεζες, θα είναι επιλέξιμες στο ευρωσύστημα από την κατεπίγουσα ανάγκη ε, χρωματοδότηση ρευστότητας, ό,τι αφορά την Ελλάδα για το T-Bills φαίνεται ότι συνδυάζεται ε, την πιθανή αύξηση του ανώτατου ορίου του Τιμπίλ στη συμφωνία με τους θεσμούς. Δηλαδή, αν υπάρχει, αν υπάρχει συμφωνία με τους θεσμούς θα αυξηθεί το ανώτατο όριο του Τιμπίλ, αλλιώς θα μειωθεί. Είναι, σωστή, αυτός, είναι σωστός ο σχετισμός που κάνω. Και τέλος, τελευταία ερώτηση. Την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μπράγκη ήρθε στην Επιτροπή και είπε ότι το ανώτατο όριο του, των Τιμπίλ είναι απόφαση του Eurogroup. Αλλά καθ' όλη την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλεγε ότι δεν θα πρέπει να αυξηθούν τα T-bills. Θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ποιο τελικά λαμβάνει την απόφαση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Eurogroup. Σας ευχαριστώ. Πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, ήδη ε, υπενήχθηκα την απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση. Είπα ότι όντως αυτό ισχύει, ότι δηλαδή αν μια χώρα ε, προβεί σε στάση πληρωμών, χρεοκοπήσει. Αυτό δεν έχει άμεση ε, επιρροή στις τράπεζες της. Αν οι ίδιες οι τράπεζες είναι φερέγγιες, αν δεν έχουν προστασία πληρωμών και αν έχουν ασφάλειες και εγγύσεις, είναι επιλέξιμες. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες, άσχετα με τη στάση πληρωμών της χώρας. Τώρα, η κατάσταση ε, σε ισχύει σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Μπορεί να επιδεινωθεί στη συνέχεια. Αυτό θα κρυθεί όμως ανάλογα με τις περιστάσεις. Πάντως, αυτόματη συνέπεια, αυτόματος αντίκτυπος δεν υπάρχει. Και ε, σε σχέση με το ισχύον πρόγραμμα στην Ελλάδα, έχουν απομείνει 10 δισεκατομμύρια περίπου και κάτι που έχουν προβλεφθεί για πιθανή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Αυτό όμως προϋποθέτει απόφαση του, του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM, του Σταθεροποιητικού Μηχανισμού, που θα μπορούσε να αποφασίσει να ενισχύσει την ε, κατάσταση των ελληνικών τραπεζών αν το κρίνει απαραίτητο. Υπάρχει αυτό το ποσό διαθέσιμο, αλλά θα εξαρτηθεί από την απόφαση ε, του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταθεροποιητικού Μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τα T-bills, ο πρόεδρος Δράγκη όντως είπε στην ε, συνεδρίαση που αναφέρατε, διαβάζοντας το ανακοινοθέν του 2012 το θεσμό της Τρόικας που προέβαινε σε αξιολόγηση της κατάστασης στην Ελλάδα δεδομένου της προοπτικής ε, της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Και η αξιολόγηση ήταν θετική, ότι δηλαδή υπήρχαν πολλές πιθανότητες και θετικές προοπτικές της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προγράμματος. Με βάση λοιπόν αυτή τη θετική αξιολόγηση, προσωρινά, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το ποσό των d που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά ως ασφάλειες. Και ερχόμαστε στο στην τρίτη ερώτηση. Εδώ έχουμε δύο τεινά, δύο όρια. Στο ελληνικό πρόγραμμα, στο δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα, είχαμε προβλέψει τις πηγές χρηματοδότησης για το ελληνικό κράτος. Και μία από τις πηγές χρηματοδότησης ήταν έκδοση T-bills, 50 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν το ανώτατο όριο που είχε καθορίσει το Eurogroup για την έκδοση των T-bills. Τώρα, άλλο το όριο των T-bills που γίνονται δεκτά ως ασφάλειες για να ε, ζητηθεί χρηματοδότηση από το, από το ευρωσύστημα, το Eurosystem, Αυτό είναι διαφορετικό όριο και τα τελευταία χρόνια είχαμε το 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το δεύτερο όριο. Αυτό το όριο προσωρινά αυξήθηκε το 2012 μετά την θετική αξιολόγηση που διάβασε ο πρόεδρος Ντράγκη στην Επιτροπή. Αυτό όμως είναι διαφορετικό. Υπάρχουν και τα δύο ανώτατα όρια, αλλά φορούν διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ. Ε, ε, και επίσης τα 50 δισεκατομμύρια που ήταν στο πρόγραμμα ε, χρησιμοποιήθηκαν τα 15 συγγνώμη. Αλλά δεν μπορούν να, χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιηθούν όλα ως ασφάλειες για να ε, φτάσουμε στο δεύτερο όριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα από ό,τι περιμένα και η ψηφοφορία FC θα αναβληθεί για μισή ώρα. Έχουμε λοιπόν λίγο χρονικό περιθώριο για να παραμείνουμε στα πέντε λεπτά ε, για ερωταπαντήσεις. Μάρκο Τσάνι για το EFTD τώρα. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ερωτήσεις για τον ε, Αντιπρόεδρο. Πρώτα απ' όλα για την διαφάνεια της ΕΚΤ και το, την πάσα που κάνατε στην εισαγωγική σας ομιλία ήταν ότι η διαφάνεια είναι κάτι που θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο και να είμαστε ικανοποιημένοι. Κάτι λοιπόν που ρώτησα και στον κύριο Ντράγκη την τελευταία φορά και δεν μου απάντησε. Δεν, εάν είναι αρμοδιότητά σας η, διαφάνεια δεν πρέπει να υπάρχουν μελέτες που να δημοσιοποιούνται για τον αντίκτυπο των νομισματικών πολιτικών ιδίω αυτών των έκτακτων μέτρων της ΕΚΤ στο ε, ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή τι ωφέλει έχει η πολιτική τη ΕΚΤ, στι ιδιωτικέ τράπεζε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ούτω καθεξή. Κρίνοντα από τα τριμηνιαία αποτελέσματα των μεγαλύτερων τουλάχιστον χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων, βλέπουμε ότι αντίκτυπο προκύπτει. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια για όλου του πολίτε και σε αυτό το σκέλο. Ε, δεύτερο σημείο. Ε, έχουμε μία ανάγκη να αξιολογήσουμε την δραστηριότητά σας ως τώρα στην TLTRO. Για τα μακροπρόθεσμα στοιχεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά από τις τράπεζες για να μπορούν να χρηματοδοτούνται και οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάμε για στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Δηλαδή, ε, αποτίμηση της ε, λειτουργίας αυτών των 200 δις που δόθηκαν στις ε, τράπεζες με το σκοπό αυτό πρέπει να γίνει. Και με ένα τελευταίο σχόλιο για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Πιστεύετε ότι όντως ένας χρηματοπιστωτικός διάβλος όπως αυτός των ε, κεφαλαγορών μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά έτσι στην Ευρώπη. Ας δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Ας το θεωρήσουμε αυτό ένα θετικό παράδειγμα. Όμως ε, το επιχειρηματικό και βιομηχανικό μοντέλο των ε, είναι πολύ διαφορετικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κίνδυνος χρηματοπιστωτικής μετατροπής των σχέσεων των τραπεζών με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στο κάτω-κάτω είναι το βασικό σκέλος τη ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι δύσκολο οι φορεί των κεφαλαίων που αν αναλύουν κυρίως τα αριθμητικά στοιχεία να αξιολογήσουν ε, την πιθανή κερδοφορία μικρών επιχειρηματικών εγχειρημάτων ή του ε, επιχειρηματικού μοντέλου της Ευρώπης που πολλές φορές αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις στη βάση του και στον ιστό του με λιγότερους από 10 εργαζομένους. Μιλάμε για στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο να τα υπολογίσει κανείς και τελικά δεν θα χρηματοδοτούνται. Και τώρα έχουμε ένα λεπτό και 20 δεύτερα για τις απαντήσεις. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα μόνο. Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να προσπαθήσω να κάνω την μπορώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, ναι. Η ανάλυση του αντικτύπου γίνεται σε, διάφορα έγγραφα εργασίας και σε διάφορα κείμενα. Θα μπορούσα λοιπόν να σας δώσω κάποιο υλικό για τον αντίκτυπο αυτό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο τραπεζικό σύστημα όλο ιδιαίτερες. Να σας πω ότι οι πολιτικές μας έχουν συμβάλει στη μείωση κατά πολύ του κόστους χρηματοδότησης για τις τράπεζες που έχει μειωθεί και ως εκ τούτου από πέρσι, στα τέλη του έτους, τα ποσοστά δανεισμού των τραπεζών και στα νοικοκυριά και στις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείε έχουν μειωθεί Συμβαίνει λοιπόν αυτό τώρα και οι δύο, και τα δύο ποσοστά μειώνονται. Οι πολιτικές μας δε δεν έχουν ως βασικό στόχο τον πληθυρισμό και την σταθεροποίηση των τιμών και στις δύο κατευθύνσεις στην Ευρωζώνη και ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί ένα κανάλι διάδοσης των πολιτικών, δεν, δεν αποτελεί τον στόχο των πολιτικών. Στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών προς αμφότερες τις πλευρές. Σε ό,τι αφορά το TLDRO, τις στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, στα τέλη του 11 και στις αρχές του 12, ήταν ε, δύο επιχειρήσεις μία στιγμή, σε μία στιγμή που οι επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση των τραπεζών είχαν λίγο πολύ παγώσει. Είχε αποτελέσματα λοιπόν το σύστημα. Και μετά από χρονικό διάστημα, όταν άλλαξε η κατάσταση, άρχισαν να ανταποδίδουν τα δάνεια οι τράπεζε. Αυτή τη φορά οι πράξει σε μακροπρόθεσμα χρηματοδότηση συνδέονται με τη συμπεριφορά σε περίπτωση πίστοση. Αυτό τι σημαίνει ότι η διευκόλυνση ισχύει για τέσσερα χρόνια, αλλά θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για την πίστοση. Ιδάλλως μετά από δύο χρόνια θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα. Δεν μπορούν να τα κρατήσουν δηλαδή για το διάστημα των τεσσάρων ετών. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η συνάρτηση με τη συμπεριφορά του της πίστοσης. Καταρχάς δηλαδή οι προϋποθέσεις για την έναρξη του προγράμματος και μετά από δύο έτη που και πάλι κρίνεται βάσει της συμπεριφοράς τους. Υπάρχει αυτή η ρεσιμότητα, πολύ σημαντική για τις ε, κεφαλικές αγορές τώρα, σε σύγκριση με τις κάνετε αυτή τη σύγκριση με την ΣΥΠΑ. Και τα δύο συστήματα μπορεί να έχουν αποτελέσματα συγκρίνοντα τι γίνεται στη ΣΥΠΑ, τι γίνεται στη Γερμανία. Δύο επιτυχεί ε, οικονομίε. Επιτυχεί με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Η ιδέα ότι τώρα οι αγορές κεφαλαίων θα αυξήσουν το ρόλο τους δεν απο... Α, με σταματάει ο πρόεδρος. Πολύ ωραία. Εντάξει. Είμαστε, απέχουμε παρασάγκας ακόμα. Έχουμε ακόμα δύο τρίτα χρηματοδότησης από τις τράπεζες στην Ευρώπη. Ε, είμαστε πολύ μακριά από την κατάσταση που υπήρχε στη ΣΥΠΑ, όπου το 20% χρηματοδοτείται από τις, μόνο από τις τράπεζες. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, επειδή παρά το γεγονός ότι έχουμε πιο πολύ χρόνο, αν οι ερωτήσεις διαρκούν 2,5 λεπτά, δεν θα ολοκληρώσουμε ποτέ στο χρονικό διάστημα των 5 λεπτών. Σας παρακαλώ λοιπόν να καταθέτω το χρονικό όριο. Μπερνάτ, μόνο. Oui, bonjour, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, τον περασμένο Μάρτιο ο κύριος Ντράγκη μου απαντούσε ότι βάσει της ΦΙΤΣ οι δράσεις της εκθερούνται θεωρούνται απόλυτα ασφαλής και ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με την πώληση ομολόγων από την πλευρά σας. Όμω, να σα θυμίσω ότι την, πτώχευση, την μέρα τη πτώχευση τη ε, Lehman Brothers ε, υπήρχε μια αντίθετη βαθμολόγηση από του οίκου αξιολόγηση διεθνώ. Ε, γι' αυτό ε, ε πρέπει να σα πω ότι την έκθεσή σα την έλαβα πολύ αργά και δεν πρόλαβα να εμβαθύνω στι λεπτομέρειε. Όμω, δεδομένων των εξελίξεων για το πρόβλημα τη ε, δευτερογενού τη αγορά, τη τραπεζική αγορά. Για το shadow banking, λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό υπάρχει για όλου του μεγάλου τραπεζικού ομίλου με ένα μεγάλο ποσοστό ποσοστών και λογον με ένα δεύτερο νόμισμα παράλληλο από το ευρώ που κυκλοφορεί στην ουσία. Αυτή την ε, προοπτική την επιβεβαιώνει και ο καθηγητή Περότη του Ιδρύματο του Άμστερνταμ καθώ και ο κύριο Σίγκε του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Τι κάνει γι' αυτό η ΕΚΤ και τι κάνουν οι υπόλοιπε κεντρικέ τράπεζε, τι κάνουν ε, για τους ε, τίτλους αυτούς που ουσιαστικά υποκαθιστούν το πραγματικό νόμισμα. Δεν υπάρχει μια, ένας ε, υπερτροφισμός εδώ που απειλεί το εθνικό νόμισμα και την ε, τραπεζική μας φερεγγιότητα. Άλλωστε η Τρόικα έχει προβλέψει την ένωση των τραπεζών και τον ενίο μηχανισμό εξυγίανσης κατά την απόψή μου. Το Front National θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές ε, αμφισημίες στα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κεντρική Τράπεζα. Ε, όσα ήδη έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για να ενισχύσει το ευρώ φαίνεται τελικά να το απειλούν ε, με το παράλληλο νόμισμα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή λοιπόν είναι εξέλιξη δράση που θα λειτουργήσει. Και έπειτα η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την επαναγορά τίτλων. Με την επαναγορά των σταθερών τίτλων που δεν του χρησιμοποιείται πλέον ω εγγύσει, ε, τι θα γίνει, τα, τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού θα εμφανίζονται στον ισολογισμό τη ΕΚΤ και όχι εκτό. Οπότε δεν πιστεύετε ότι έτσι θα αυξηθεί ο συλλογισμό τη, ε, τα αποτελέσματα θα αυξηθούν για την ΕΚΤ μέχρι το τέλο του 2016. Κωνσταντσιο, ευχαριστώ για τι ερωτήσεις σα, Ό,τι αφορά τι εξελίξει για τον ρόλο των χρηματαγορών στην χρηματοδότηση τη οικονομία, όπω έχω ξαναπεί, στην Ευρώπη, έχουμε μια οικονομία βασισμένη στι τράπεζε. Δύο τρίτα τη χρηματοδότηση τη οικονομία βασίζονται στι τραπεζικέ ενέργειε και μόνο τα υπόλοιπα στις ε, χρηματαγορές. Τελείως διαφορετικά από ό,τι στις είπα, όπου οι τράπεζες ε, μόνο το 20% της πραγματικής οικονομίας, των απαιτήσεων τέλος πάντων της οικονομίας καλύπτουν. Αυτός ο ρόλος των ε, χρηματαγορών είναι κάτι γνωστό και υπάρξει τέτοιων τίτλων. Δεν υποκαθιστούν κανένα πραγματικό νόμισμα. Μιλάμε για αξιόγραφα που εκφράζονται το σε σε ευρώ δεν υπάρχει άλλο παράλληλο νόμισμα. Και επειδή αυτά τα αξιόγραφα, αυτοί οι τίτλοι ε, ενέχουν έναν βαθμό κινδύνου και πιστοτικό και απόδοση όταν είναι υψηλότερο επίπεδο ρήμανση, δεν ε, υποκαθιστούν το χρήμα, δεν έχουν το βαθμό ρευστότητα που μπορεί να έχει το πραγματικό χρήμα. Οπότε να μην τα μπερδεύουμε. Οι εξελίξεις αυτές στον ρόλο των ιδρυμάτων, ε, των τραπεζικών ιδρυμάτων και των χρηματαγορών όντως λαμβάνουν χώρα και εξελίσσονται ε, σε ένα μέρος του χρηματοοικονομικού τομέα που είναι εξωτραπεζικός. Συμβαίνει αυτό. Έχουμε ήδη επισημάνει, όχι μόνο εμείς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα ιδρύματα, ε, έχουμε επισημάνει ότι η διόγκωση αυτού του νέου τμήματος του χρηματοπιστωτικού συστήματος πρέπει να ε, γίνει αντικείμενο αποπτίας κάποια στιγμή. Διότι αρχίζουν να προκύπτουν νέοι, νέα είδη κινδύνου Καινούριε απειλές. Αυτό το παρακολουθούμε λοιπόν στενότατα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιοι είναι αυτοί κίνδυνοι τώρα. Είναι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα και την ε, μετατροπή. Τα ιδρύματα που λειτουργούν στις κεφαλαιαγορές και την χρηματοδότησή τους έχουν χαμηλότερη μόχλευση από ό,τι τράπεζες. Διότι κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται με την έκδοση ανανεώσιμου κεφαλαίου και όχι με καταθέσει και τέτοιες είδους εγγύσεων. Άρα η μετατροπή της ορίμανσης ή της ρευστότητας είναι κίνδυνος που αφορά περισσότερο αυτές τις νέες πτυχές. Και χρειάζονται και νέα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Το έχω αναφέρει σε πολλές από τις ομιλίες μου, το έχω αναφέρει και άλλοι συναδελφοί μου. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με παράλληλα νομίσματα, όπως είπατε, που υποκαθιστούν ή διαβρώνουν το όλο σύστημα. Και στην τελευταία σας ερώτηση, πολύ σύντομα, αξίζει τα αποτελέσματα, διόγκως τα αποτελέσματά μας, ε, το εξηγήσαμε, προβλέπαμε ότι τα 60 δις των εξεγράφων που θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε μπορούν να μας φτάσουν σε αποτελέσματα που είχαμε την άνοιξη του 2012, αλλά όχι παραπάνω. Για τώρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ πέρα, κυρία Hübner. Θυμάμαι τι εποχέ ε, που θέταμε τα θεμέλια ε, εδώ για τον νέο επιπτωτικό μηχανισμό. Χαίρομαι που σα ξαναβλέπω εδώ. Θα ήθελα να σα ρωτήσω για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Γιατί μου κάνει εντύπωση που δεν είχα ακούσει ποτέ τέτοια έντονη κριτική για την Ένωση αυτή όπως αυτή που ακούω από εσάς τώρα. Λέτε ότι πλήρης ε, ρυθμιστική εναρμόνιση είναι προϋπόθεση. Από τον Επίτροπο ακούμε όμως ότι θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία αυτή. Δεν πρόκειται για μια σύντομη διαδικασία, αλλά για μια μακροπρόθεσμη και για μια αλλαγή που θα προέλθει και από την νομοθεσία αλλά και από τις ίδιες τις αγορές. Αναρωτιέμαι λοιπόν, υπάρχει μήπως μια διαφορετική κατηγορία στοιχείων, αν ε, πρέπει να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερη ερώτηση. Εσείς ως ΕΚΤ ε, έπρεπε να καταλήξετε, να, να χρησιμοποιήσετε, αναγκαστήκατε να χρησιμοποιήσετε έκτακτα μέτρα. Μήπως αυτό το αποτελεί πλέον το new normal, ε, την, τη νέα κανονική κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, για την υπενθύμηση, της κοινή μα δουλειά κατά το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την ε, Ένωση Κεφαλαγόρων, προσπάθησα να υπογραμμίσω την ανάγκη να μην ξεχάσουμε τη φιλοδοξία του project. Είμαι απόλυτα, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι δεν μπορεί αυτό να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι αλήθεια και υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή που είναι πιο απλά και θα πρέπει να αποτελέσουν τα στοιχεία με τα οποία θα ξεκινήσουμε. Όπως για παράδειγμα, επιμένουμε με την Τράπεζα της Αγγλίας στο ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί ένας νέος τύπος απλών και διαφανών Αυτό αποτελεί τμήμα της χρηματοδότησης που αποτελεί τμήμα της Ένωσης Κεφαλαγορών. Αποτελεί λοιπόν ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στο, στην πράσινη βίβλο της Επιτροπής. Είναι ένα στοιχείο. Αλλά προσπάθησα και πιστεύω ότι η ΕΚΤ και το σύστημα της Ευρωζώνης θα ακολουθήσουν τις ίδιες γραμμές να πω ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε τον απότερο στόχο της ε, Ένωσης Κεφαλαγόρων και αυτό ε, συμπεριλαμβάνει και μια μεγάλη προσπάθεια, ένα μεγάλο εγχείρημα Η Ιδάλλως δεν μπορούμε να μιλάμε για ένωση υπό την κανονική ένωση. έννοια. Ας μην ικανοποιηθούμε και αρκεστούμε σε κάποια μικρά επιτεύγματα που μπορούν να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα. Να μην χάσουμε από το στόχαστρο του πιο φιλόδοξους στόχους της Ένωσης Κεφαλαγορών. Υπό αυτή την έννοια μίλησα. Δεύτερη ερώτηση για τα μη τυποποιημένα μέτρα. Όχι, δεν αποτελούν το καινούριο κριτήριο, το new normal. Δεν υπάρχει πρόθεση να συνεχίσουν. Βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση πολύ χαμηλού πληθωρισμού. Ελπίζουμε αυτό να διορθωθεί. Γιατί υπάρχουν και κίνδυνοι στην κατάσταση αυτή, στην κατάσταση αυτή σε ό,τι αφορά τον χαμηλό πληθωρισμό. Ε, αυτό είναι κακό για την οικονομία για διάφορους λόγους. Ελπίζουμε λοιπόν να εξέλθουμε από την κατάσταση αυτή και όταν εξέλθουμε από την κατάσταση θα πάψει και η χρήση των μέτρων αυτών. Και οι κεντρικές ε, τράπεζες θα επιτρέψουν στην νομισματική πολιτική και τα κανονικά επιτοκία για τη διαχείριση της οικονομίας. Όχι, δεν πρόκειται για ένα new normal. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες το λόγο έχει ο συνάδελφος Άλβαρες. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ θα υποβάλλω και πάλι ερωτήσεις για αυτό το σχέδιο της ε, Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών, CMU και τη σχέση που έχει με τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στον εποπτικό ρόλο που πρόσφατα ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, επί των τραπεζών στα πλαίσια της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Εστεριζόμαστε το στόχο της βελτίωσης κατάστασης στον τραπεζικό κλάδο, αλλά η αύξηση της χρηματοδότησης μέσω μη τραπεζικών φορέων ίσως δημιουργήσει προβλήματα αν δεν εξασφαλιστεί πανευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός, κάτι που είδαμε ότι συνέβη με τις τράπεζες στην τελευταία κρίση. Πώς βλέπετε λοιπόν τον εποπτικό σας ρόλο, τις εποπτικές σας δραστηριότητες Χρειάζεται ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο και ένα κοινό υποπτικό πλαίσιο για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Επίσης, ε, είπατε ότι για να... η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών θα βελτιώσει την ε, νομισματική πολιτική, αλλά η νομισματική πολιτική ε, κυρίως εφαρμόζεται από τα τραπεζικά ιδρύματα. Πώς λοιπόν βλέπετε αυτή την καλύτερη διαβίβαση ή μεταβίβαση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Πολιτικής μέσω της Ένωσης Κεφαλαγορών. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Είπα στις αγωγικές μου παρατηρήσεις ότι η Ένωση Κεφαλαγορών έχει πολλά πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα αυξάνει την διασύνδεση και την αλληλεπίδραση των ε, χρηματοπιστωτικών συστημάτων και μάλιστα με πιο έντονο τρόπο και ίσως αυξήσει τον κίνδυνο της μετάδοσης αν ε, λάβει χώρα κάποιο ατύχημα σε κάποιο σημείο του συστήματος εξαιτία τη ενισχυμένη αλληλεπίδραση. Οπότε η Ένωση Κεφαλαγορών όπω και η Τραπεζική Ένωση σημαίνουν ε, ανάγκη διευρυμένου εποπτικού μηχανισμού και εξασφάλιση συνθήκων ισότιμου ανταγωνισμού για να αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι της ε, μετάδοσης των ατυχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι ε, οι φορείς, μιλούμε για χρηματαγορές, κεφαλαγορές, ε, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την, ε, για, την εποπτεία θα πρέπει να ενισχύσουν το ρόλο τους. Και μακροπρόθεσμα, σε τελική ανάλυση και όταν εφαρμοστεί πλήρωση όλη η διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι κάποια στοιχεία εποπτείας θα πρέπει να μεταφερθούν, να εκχωρηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Τραπεζικής Ένωσης. Ίσως όχι αμέσως, αλλά μακροπρόθεσμα, ακριβώς για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη εποπτεία της κατάστασης και να αποφευθούν οι κίνδυνοι μετάδοσης. Επίσης, να εξασφαλίσουμε το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και ένα και συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική, θα ήθελα η συντομία να πω ότι ε, πώς διευκολύνεται από την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Καταρχήν, μια και οι συνομιλητές μας εδώ είναι οι τράπεζες, ό,τι αφορά την παροχή ρευστότητας ή την, τον άμεσο αντίκτυπο στην πολιτική των επιτοκίων. Είναι σημαντικό α, ε, αυτό το να μεταφέρεται σε όλη την καμπύλη των διαφορετικών λεξιπρόθεσμων ομολόγων. Και αυτό είναι ο ρόλο των κεφαλαιογορών, να γίνεται σωστή μετάδοση και άλλων ε, μέσων των ε, ε, αποτελεσμάτων των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Γιατί η νομισματική πολιτική μόνο τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια επηρεάζει. Και ανάλογα με το έργο των χρηματαγορών, των κεφαλαγορών, αυτά τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια μεταφέρονται και σε άλλα επίπεδα ε, τίτλων που έχουν μεγαλύτερη περίοδο λικτότητας και που είναι σημαντικά για Μακροπρόθεσμε επενδυτικέ αποφάσει γιατί δεν είναι τα εβδομαδιαία ή τα μηνιαία επιτόκια που είναι σημαντικά για τι επενδύσει, αλλά τα πιο μακροπρόθεσμα επιτόκια, γιατί οι επενδυτικέ αποφάσεις αφορούν πενταετία-δεκαετία. Οπότε εκεί διευκολύνουν το έργο οι κεφαλαγορέ, γιατί είναι πιο βαθίε αγορέ, με μεγαλύτερη ρευστότητα, έτσι ε, εξασφαλίζεται χάρη στην Ένωση Κεφαλαγορών καλύτερη μεταβίβαση τη νομισματική πολιτική. Ο κύριο Κίρτσος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω δύο ερωτήσεις. Το θέμα είναι, το, η πρώτη έχει σχέση με τα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει πολύ δυναμικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους του χρήματος. Ήθελα να ξέρω όμως, είστε ικανοποιημένος, περνάει αυτό το, η μείωση του κόστου του χρήματος στις επιχειρήσεις στο βαθμό που πρέπει να περνάει ή για παράδειγμα οι ανάγκες του τραπεζικού συστήματος εμποδίζουν ε, να περάσει το σύνολο του, της μείωσης του κόστου του χρήματος, γιατί και οι τράπεζες θέλουν την κερδοφορία τους, έχουν τη στρατηγική τους. Μήπως συγκρούεται σε αυτή τη φάση η, στρατηγική των τραπεζών με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και ποια, είναι η εκτίμησή σας και ποιος είναι ο ρόλος σας ε, σε αυτό το θέμα. Και μετά ήθελα για το Capital Markets Union που υποθέτω ότι αποτελεί ένα πλεονέκτημα των, ε, των Αμερικανών σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Ε, αυτό είναι, αν έχετε μια συνολική εικόνα των πολιτικών, οικονομικών, διαδικαστικών δυσκολιών. Άρα μιλάμε για κάτι που μπορεί να συμβεί σε δύο χρόνια, σε τέσσερα χρόνια, σε έξι χρόνια. Πότε μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Well, uh, thank you. Uh. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ναι, τα επιτόκια σε όλες τις αγορές ε, πέφτουν. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αγορά τραπεζικών δανείων. Πολύ σημαντικός κλάδος για μια περίοδο το 2012 και 2013 οι πολιτικές μας επηρέασαν τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών. Το κόστος όμως του δανεισμού από τις τράπεζες δεν ε, κινήθηκε αναλόγως. Τώρα λοιπόν αυτό συμβαίνει πλέον. Τα επιτόκια έπεσαν για τις ε, ε, επιχειρηματικές, επιχειρηματικά ομόλογα. αυξήθηκαν 13% κατά 13% τα equities από την απόφαση μας τον Γενάρη. Το κόστος δηλαδή των μετοχών μεταβλήθηκε και παράλληλα μειώθηκαν και τα επιτόκια. Να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Αυτά είναι κατά μέσο όρο. Κατά μέσο όρο. Επιτόκια σε μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 2,34% σήμερα. Ενώ το καλοκαίρι του περσινού έτους είμαστε 16 ποσοστίες μονάδες παραπάνω κατά μέσο όρο απόδοση των ε, corporate bonds 2%, το κόστος των αξιγράφων 7%, επίπεδο αντίστοιχο με αυτό που ήταν πριν από την κρίση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του spillover, της διάδοσης της πολιτικής μας και σε άλλες αγορές. Αυτό μειώνει το κόστος κεφαλαίου και για, με τις, για τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά τις επενδυτικές αποφάσεις και την περαιτέρω ανάπτυξη. Η δεύτερη ερώτηση. Θα είναι μακρά διαδικασία, σίγουρα. Είναι δύσκολη, είναι ευαίσθητη. Πιστεύω όμως ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορούν να συγκριθούν οι προσπάθειες που έγιναν κατά τα παρελθόν στην Ευρώπη και απέτυχαν. Υπήρχαν κάποιες απόπειρες εναρμόνισης του εταιρικού δικαίου, συζήτησης κάποιων τέτοιων πτυχών πλέον ε, με την κρίση πίσω μας. Το project της Τραπεζικής Ένωσης έχουμε κάποιες ε, πολύ τολμηρές αποφάσεις θεσμικής φύσης που ήταν απαραίτητες και θεωρώ ότι και αυτές θα συμβάλλουν εν ευθέτω χρόνο και θα μιλήσουμε υπέρ των πλεονεκτημάτων και των όφελων των πρωτοβουλίων αυτών. Να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι να μην βρεθούμε σε μία δομή όπου οι τράπεζες θα χρηματοδοτούν μόνο κατά 20%. Όχι. Η Ευρώπη και οι επιτυχείς χώρες στην Ευρώπη έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά χωρίς μια τέτοια δομή και πιστεύω ότι χρειάζεται μια σωστή συμμετοχή των τραπεζών σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τους σοσιαλιστέ και δημοκράτες. για καλή. Uh, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά και πάλι τα προβλήματα ρευστότητας που θα έχει ε, βρέχει πρόθεσμα η Ελλάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται ε, για το Μάιο είναι σχεδόν ένα δις ε, η ρευστότητας από την έκτη προς την Ελλάδα. Αν υπάρχει σχέδιο ποιο είναι το σχέδιο της έκτη ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες σε περίπτωση που δεν ληφθεί συμφωνία, όχι, ε, δεν ληφθεί συμφωνία, όχι σε περίπτωση τάσης πληρωμών, αλλά σε περίπτωση μη ε, συμφωνίας. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα τέτοιο πιστοτικό γεγονός, τι θα κάνει με το ELA η Ελλάδα προκειμένου να συγκρατηθεί ο συστημικός κίνδυνος στις ελληνικές τράπεζες. Θεωρεί η λαμβάνει υπόψη την δυνατότητα να επιβάλλει ελέγχους ε, δανεισμού στις ελληνικές τράπεζες και η επιβολή τέτοιων κεφαλαιακών περιορισμών δεν σημαίνει κατά ανάγκη Brexit. Και η αξία των αγγιήσεων που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες για να, να πάρουν την χρηματοδότηση από το ΕΛΑ μειώνεται. Οπότε έχουμε ένα κούρεμα ουσιαστικά των ασφαλιών. Ποιο είναι το ποσοστιαίο μέγεθος αυτών, τον, αυτού του κουρέματος σε περίπτωση ατυχούς ε, γεγονότος ενός πιστοτικού ατυχήματος. Επίσης, αν η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στην Ελλάδα είναι σταθερά στοιχεία του ενεργητικού που δεν ε, τα εγγυάται το σύστημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας τι θα γίνει σε περίπτωση πιστοτικού γεγονότος. Ε, θα μπορέσει να παραμείνει ο ελληνικό τραπεζικός κλάδος ανθεκτικό και βιώσιμος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ήδη προανέφερα ότι οι κανόνες που ισχύουν για την παροχή ρευστότητα στι τράπεζες εξαρτώνται από το κατά πόσο είναι φερέγγιε, από το κατά πόσο έχουν αξιολογηθεί ως φερέγγιε και αν έχουν επιλέξει με ασφάλειες και εγγύησεις για να λάβουν τη χρηματοδότηση αυτή. Και αυτό ισχύει και για το ELA, την έκτακτη αυτή χρηματοπιστωτική γραμμή. Το ELA ισχύει και για τα δύο. Οπότε, αν δεν έχουμε ασφάλειες, δεν έχουμε εγγύσεις, δεν δώσουν οι τράπεζες εγγύσεις. φυσικά δεν είναι επιλέξιμες για την παροχή λευστότητας χωρίς παροχή εγγύσεων. Οπότε οι τράπεζες θα χρειαστεί να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους τη αυτή περιπτώσει. περίπτωση. Απευχόμαστε βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά αυτά προβλέπουν οι κανόνες. Επίσης, όπως προανέφερα, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, όπως έχει προταθεί και όπως έχει εγκρίνει και το Διοικητικό του Συμβούλιο, ε, οι ελληνικέ τράπεζε θα πρέπει να αυξήσουν την έκθεσή του προ το κράτο, προ τα κρατικά ομόλογα, ώστε να μην γίνουν ακόμη περισσότερο εξαρτημένε ε, σε περίπτωση πιστοτικού γεγονότος ε, τη χώρα. Αυτό ήταν και το σκεπτικό τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε αν λάβει χώρα στάση, στάση πληρωμών, η συνθήκη όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν προβλέπει μια χώρα που προβαίνει σε στάση πληρωμών να αποπευθεί από την Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Οι συνθήκες δεν προβλέπουν τέτοια δυνατότητα από αποπομπής μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Και οι, οι τράπεζες ε, υπάγονται στους κανόνες και αντιμετωπίζονται ανάλογα με τους κανόνες. Τώρα, σε σχέση με το προηγούμενο το ισχύον πρόγραμμα, έχουμε πάνω από 10 δισεκατομμύρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αν παραστεί ανάγκη, κάτι που δεν ισχύει τώρα. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, ανάλογα με τις περιστάσεις, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, αλλά από τους υπουργού ΕΚΟΦΗΝ και όχι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε, εμείς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το μόνο που μπορεί να πει είναι εφαρμογή των κανόνων, όπως σας είπα. Δεν μπορούμε εμείς να υποβάλουμε σχέδια οι προτάσεις. Και η ασφάλεια, η παροχή εγγύσεων από τι τράπεζες είναι σημαντική. Αναφερθήκατε σε ε, ελέγχους κεφαλαίων και δανεισμού. Οι έλεγχοι, οι έλεγχοι κεφαλαίων ε, θα επιβληθούν μόνο εφόσον το ζητήσει η, Ευρωπαϊ... η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί η, η απόφαση αυτή να ληφθεί έξωθεν της Ελλάδας. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να το ζητήσει και ε, επιπλέον, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει την πρόταση. Πάντως, το αρχικό αίτημα θα πρέπει να προέλθει από την ελληνική κυβέρνηση. Και όπως είδαμε και στην περίπτωση της Κύπρου, οι έλεγχοι κεφαλαίου δεν οδήγησαν σε έξοδο από το ευρώ, σε έξοδο από την ευρωζώνη. Η Κύπρος ε, τελικά ε, ε επιτυχώς ολοκλήρωσε και θέσε τέρμα στους ελέγχους κεφαλαίων και παρέμεινε στην Ευρωζώνη παρά την εφαρμογή αυτών των ελέγχων κεφαλαίου και σταδιακά τους κατήργησε όσο αυξανόταν η εμπιστοσύνη και ολοσχερός τους εξάλληψε τελικά. Οι τρεις τελευταίοι ομιλητές, τρία λεπτά για να μπορέσουμε να έχουμε τις ψηφοφορίες. Σίκπιτ Μούνεσαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διπρόεδρε, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξηγήσει αυτές που μας δώσατε. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό και σε ό,τι αφορά το, τις θετικές επιπτώσεις της προσωπικής χαλάρωσης. Ανησυχώ για τους ενδεχόμενους κινδύνους, ωστόσο, που διαγράφονται. Ένας εξ αυτών είναι ε, ο ισολογισμός του ιδιωτικού τομέα λόγω της συνεχιζόμενης μη απόδοσης συγκεκριμένων στοιχείων και λόγω της μεγάλης χρέωσης ε, του, δημόσιου, του ιδιωτικού κλάδου σε κάποιες χώρες. Αυτό φυσικά οδηγεί σε μεγάλη εξάρτηση. Ρωτώ λοιπόν, η ΕΚΤ τι θέλει να κάνει για να αντισταθμίσει αυτές τις τάσεις, αυτό είναι το πρώτο θέμα και το δεύτερο θέμα που έχω να θέσω ένα άλλο πρόβλημα για την προσωπική χαλάρωση είναι η κατάσταση με τους θεσμικούς επενδυτές. Ε, τα συνταξιδευτικά ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται σε μια δύναμη θέση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και σε ό,τι αφορά το μηχανισμό προσωπική χαλάρωση και τη μετάδοση, διάδοση τη προσωπική χαλάρωση. Τι θα κάνει λοιπόν η ΕΚΤ για να διασφαλίσει ότι η ανάληψη ρίσκου στην Ευρωζώνη θα καταστεί εκ νέου βιώσιμη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, αναφερθήκατε στην κατάσταση σε ό,τι αφορά την υψηλή χρέωση και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη. Η πολιτική όμως ε, της επικρατικής ε, νομισματικής πολιτικής που μειώνει τα επιτόκια βοηθά την κατάσταση αυτή γιατί μειώνεται το βάρος του χρέους. Άρα αντί να αυξάνουμε το ρίσκο και τον κίνδυνο σε ό,τι αφορά τις χρεωμένες, τα χρεωμένα θεσμικά όργανα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε προκειμένου να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος του χρέους και ελπίζουμε σε βάθος χρόνου να μειώσουν το ποσοστό χρέωσης και εδώ χρειάζεται η μόχλευση όντως, αλλά εδώ πέρα δεν αυξάνουμε τους κινδύνους σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους θεσμικούς επενδυτές. Διαφέρει η κατάσταση ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο των θεσμικών οργάνων. Μίλησα ήδη πολύ για τους ασφαλιστές και όντως οι ασφαλιστές είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην κατάσταση με τα κέρδη που σημείωσαν μέσω αύξησης των τιμών των στοιχείων. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους και τις υποσχέσεις για απόδοση στο νέο περιβάλλον θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες σε μια κατάσταση χαμηλών επιτοκίων. Ευχαριστώ. Ο Κώστας Μαυρίδης για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Right here. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Θα μιλήσω ελληνικά. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Are you listening? Uh, Capital Market Union. Η αγορά, η Ένωση Κεφαλαίων Αγορών. Δύο γεγονότα. 13 ε, εκατομμύρια ευρώ είναι σε savings bank accounts. Και το δεύτερο γεγονός, έχουμε μια τεμαχισμένη αγορά, fragmented market. We all agree on that. Τι νομίζετε θα μπορούσε να βοηθήσει τεχνοκρατικά και όχι πολιτικά να σταματήσει αυτό το, η έξοδος κεφαλαίων από τις χώρες της περιφέρεια, Ευρωπαϊκής Περιφέρειας να κινηθούν, να έχουμε μια καλύτερη μακροοικονομική ισορροπία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα επιτόκια, για το κόστος άντλησης κεφαλαίων των τραπεζών και όλα αυτά. Δεύτερο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, to transform ELA, e, ε, Emergency Liquidity Assistance, into long-term bonds. Θα το μελετούσατε αυτό για μια περίπτωση μιας τράπεζας, για παράδειγμα, η οποία έχει επανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως. Και το τρίτο, της προάλλες, επειδή αναφερθήκατε στην περίπτωση της Κύπρου, τις προάλλες στην Κύπρο πέρασε το τελευταίο η νομοθεσία για αφαιρεγκαιότητα. Ήθελα να ξέρω, η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την ποσοτική χαλάρωση. Σας ευχαριστώ. Ε, thank ε, Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορώ για την έξοδο κεφαλαίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και κάθε χώρα, βασίζεται σε, μια, σε βασικές ελευθερίες. Και μία από αυτές είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτήν την έννοια, οποιοδήποτε περιορισμός του διοικητικού ελέγχου μπορεί να είναι έκτακτη μόνο κατάσταση, όπως έγινε στην Κύπρο. Η κανονική κατάσταση είναι ότι είναι απόλυτα ελεύθερη η κυκλοφορία των κεφαλαίων για τους πολίτες και τις εταιρείε σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν υπάρχει λοιπόν όταν υπάρχει έξοδος κεφαλαίων είναι μια τάση των νεοκαιριών, των ιδιωτών και των εταιριών όταν βλέπουν ένα κίνδυνο ε, οικονομικό κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν κίνητρο να μετακινηθούν, να μετακινηθούν τα κεφαλαία τους εκτός του, της περιοχής κινδύνου. Εάν λοιπόν θέλετε εξήγηση για το λόγο για τον οποίο η Ελλάδα ε, έζησε τέτοια έξοδο κεφαλαίων από τον Δεκέμβριο, αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική κατάσταση και τις πολιτικές αποφάσεις της Ελλάδας. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Το γεγονός ότι ως τώρα δεν επετέχθη συμφωνία με τα άλλα κράτη-μέλη ήδη σημαίνει πολλά. Αυτό δημιουργεί βεβαιότητα και γι' αυτό υπάρχει έξοδος. Ο μόνος λόγος να αντιμετωπιστεί αυτό είναι να εργαστούμε προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με τα υπόλοιπα κρατημέλη. Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας. Σε ό,τι αφορά το ELA και την μετατροπή του σε μακροπρόθεσμα ομόλογα, αυτό είναι εκτός των κανόνων μας. Ευχαριστώ. Τελευταίος σε τον κατάλογο ο Τόμας Μάνια, το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κωνσταντσιό, θα πρέπει να ξαναθέσω το θέμα του χαμηλού επιτοκίου που επικρατεί. Οι επενδύσεις ε, και οι εμπιστοτές ε, αρέσκονται σε αυτά, αλλά όχι οι υπόλοιποι. Ε, στη Γερμανία έχουμε απώλεια τα τελευταία πέντε χρόνια στους αποτεμιευτές 190 δισεκατομμύρια ευρώ αυτό δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Η Σιλβί Γκουλάγα δικαίω ε, ε, επεσήμενε τι γίνεται με τι ε, ασφαλίσεις ζωή. Και επίση τα συνταξιδοτικά ταμεία. Υποσχεθήκαμε 3,5 έω 4%. Αυτά ήταν η εγγύηση. Η εγγύηση είναι ένα μέτρο για την οικοδόμηση, οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Όχι κάτι με το οποίο παίζουμε. Είπατε ότι πρέπει να υπάρξει προσαρμογή. Ναι, για το μέλλον. Αλλά τι θα γίνει με τις δεσμεύσεις που έχουμε ήδη αναλάβει. Και πέρα από τις επιχειρηματικές συντάξεις, το γενικότερο κλίμα, οι ιδιωτικές ασφάλειες, οι ιδιωτικές συντάξεις. Πώς μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα ασφαλές ε, ποσοστό. Δεν είναι μόνο πολιτικό και χρηματοπιστωτικό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας να ξεκινήσω επισημένοντά το εξή. Να σας αναφέρω ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε στο οικονομικό δελτίο τη Γερμανικής Κεντρική Τράπεζας πριν από κάποιου μήνες, όπου κατέδειξαν ότι σε πραγματικούς όρους, σε πραγματικούς όρους αυτό έχει σημασία. Τα επιτόκια των καταθέσεων στη Γερμανία σήμερα είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν το 2006 και το 2007. Τότε τα επιτόκια στις καταθέσεις, κανονικές καταθέσεις, ήταν στο 2,6%. Ο πληθωρισμός όμως ήταν επίσης στο 2,6%. Άρα μηδενική μηδενικό το αποτέλεσμα. Τώρα ο πληθωρισμός στη Γερμανία είναι στη μισή ποσοστία μονάδα. Οι καταθέσεις ε, λοιπόν συνδέονται με τι πληθωρισμό αυτό. Πάλι μηδενικό λοιπόν, μηδενική σχέση. Αυτό το αμελούμε, γιατί φυσικά ο κόσμος έχει την τάση να σκέφτεται με ονομαστικές ε, αξίες. Έχει κάποιες τέτοιες ψευδεστήσεις. Εσείς όμως Γερμανός νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτά λόγω της κουλτούρας που επικρατεί στη Γερμανία τα θέματα χρήματων και γιατί είναι σημαντικός ο πληθωρισμός για την πραγματική αγοραστική δύναμη. Τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Τα επιτόκια τώρα είναι χαμηλά επειδή ο πληθωρισμός είναι πολύ χαμηλός και εργαζόμαστε με τις πολιτικές μας για να αυξήσουμε τον πληθωρισμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Όταν συμβεί αυτό, τα επιτόκια εκ νέου θα αυξηθούν. Αν υπάρξει βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας θα είναι θετικά με πραγματικούς όρους και πάλι όπως ήταν στο παρελθόν τα επιτόκια. Άρα βρισκόμαστε σε μια προσωρινή κατάσταση, οι πολιτικές μας λειτουργούν και σκοπό έχουν να διορθώσουν αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επανέλθουμε σε μια κατάσταση φυσιολογική, πιο φυσιολογική από τώρα. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι αυτά που κάνουμε προκαλούν την κατάσταση. Όχι, δεν προκαλέσαμε τον χαμηλό αυτό πληθωρισμό. Και όπως σας είπα, δεν φταίει μόνο το πετρέλαιο, γιατί και εκτός του πετρελαίου το πληθωρισμός είναι με 0,6% που και αυτό είναι πολύ πιο χαμηλό από το ποσοστό που είχαμε ως συντολή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ο Πρόεδρος, κύριε Διπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Κωνστάντσιο, για την αναλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σας για το αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ και εσάς συναδέλφοι που ολοκληρώσαμε τόσο γρήγορα. Ήταν ε, πολύ καλή η διεκπαιρέωση γιατί στις 16.45 πρέπει να γίνει η ψηφοφορία και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Φέρμπερ για τις ψηφοφορίες. Να ευχαριστήσω εκ νέου τον κύριο Κωνσταντσίου που παρευρέθηκε μαζί μας σήμερα. <laughs>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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen dann... Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Να σας παρακαλέσω να πάρετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Haben Sie alle Ihre Stimmkarte? Βάλατε όλες τις κάρτες σας παρακαλώ. Στη συσκευή. Κυρία Περές, αν μας επιτρέπετε να ψηφίσουμε... να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Δοκιμαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Δεν έχει λήξει ακόμα η ψηφοφορία, η δοκιμαστική. Όλοι οι περήφανοι κατοχοί κάρτας ψήφισαν. Πέρας της ψηφοφορίας, μάλιστα όλες οι ομάδες λοιπόν ψήφισαν. Να περάσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν για την έκθεση του συναδέλφου Μαυρίτη. Συμβιβαστική Α, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Με προφορική τροπολογία των πρασίνων. Την έχετε όλοι. Να ψηφίσουμε καταρχάς την προφορική τροπολογία των πρασίνων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του συμβιβαστική Β με την προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστή, ε, είναι 24 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Να ψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την τροπολογία 25 έναρξη ψηφοφορίας. Εάν ψήφισατε όλοι, Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία εδώ. Εγκρίνεται. Ε, επαρκή διαφορά, λέει ο πρόεδρος. Συμβιβαστική C. Α, μου είπαν από πλευράς του ΕΛΚ ότι υπάρχει έτοιμα για χωριστή ψηφοφορία. Ψηφοφορία στα τμήματα. Αληθεύει. Συμπεριλαμβάνεται αυτός ο καταλόγος ψηφοφορίας. Α, δεν το έχουν οι άλλοι. Ναι, και εγώ δεν το ήξερα. Θα μπορούσε κάποιο από το ΕΛΚ να μα παρουσιάσει πώς θέλει να γίνει η ψηφοφορία κατά τμήματα. Κύριε Μπάλτς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλαμε στην παράγραφο 3 στο κείμενο αναφέρονται το labor intensive, έντες εργασίας. Εδώ θα θέλαμε να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία το συζητήσαμε και το συμφωνήσαμε και με τις σκιώδη ηγήτρια της ομάδας μας. Μάλιστα, για το labor intensive, αυτό θέλουν να ψηφίσουν χωριστά. Να ψηφίσουμε λοιπόν καταρχάς για τη συμβαστική C χωρίς την ε, labor intensive. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής C χωρίς την διατύπωση labor intensive, παρακαλώ. Είσαστε κατά? Ναι, η ε, κυρία Φερέρα. Ναι, κοιτάξτε, ρώτησα και τους βοηθούς μου, δεν είχαμε πληροφόρηση, δεν έχουμε οτιδήποτε... Ε, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή την τροπολογία. Νομίζω ότι έτσι λοιπόν λέει ο Πρόεδρος απορρίπτεται η προφορική τροπολογία να ψηφίσουμε το σύνολο της συμβαστικής C. Υπέρ. Κατά. Η διαδικασία είναι μάλλον ε, εύκολη. Ξεκινάμε ψηφίζοντα τη συμβαστική C χωρί την διατύπωση labor intensive και μετά θα ψηφίσουμε για τις λέξει labor intensive. Εγώ θα ψήφιζα και τι δύο φορέ υπέρ. Αν ήμουν σοσιαλιστή που δεν θα σημαίνει ποτέ. Πρόεδρε, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Δεν έχουμε το κείμενο μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι ε, συμβαίνει άμα συμπεριληφθούν ή διαγραφούν αυτέ οι λέξεις labor intensive. Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται από δικαστικής άποψη. Πρέπει να το έχουμε ανακοινώσει από πριν. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε ξαφνικά σε διάφορα αποσπάσματα να, να βγάζουμε λέξει χωρίς να ξέρουν οι υπόλοιποι βουλευτές τι συνεπάγεται αυτή η αφαίρεση. Γι' αυτό είμαι αντίθετος. Ναι, κοιτάξτε συνάδελφε, έχετε μπροστά τον ε, κατάλογο της ψηφοφορία και τα συμβαστικά κείμενα τα έχετε επίσης. Θα βρείτε τη συμβαστική και εκεί θα διαπιστώσετε ότι στα αγγλικά εμφανίζεται ο όρος labor intensive για την επιλογή έργων και την πρόθεση έργων ε, έντασης εργασίας. Το ΕΛΚ θέλει να αφαιρεθεί αυτή η διατύπωση για να μην υπάρχει τέτοιος όρος για τα project. Δεν είναι προφορική τροπολογία, είναι ψηφοφορία κατά τμήματα. Αυτό πάντα έως τώρα το επιτρέπεται η διαδικασία. Το κείμενο το έχετε εδώ και καιρό μπροστά σας. Μάλιστα, πάμε πάλι. Συμβιβαστική C, χωρίς το labor intensive. Ποιος είναι υπέρ. Και οι σοσιαλιστές θα πρέπει να είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Άποχες. Άρα εγκρίνεται ο συμβιβασμό χωρί τι δύο αυτέ λέξει. Τώρα να ψηφίσουμε τι δύο αυτέ λέξει. Labor intensive. Όποιο θέλει να τι ε, συμπεριληφθούν θα ψηφίσει υπέρ. Όποιο δεν θέλει να συμπεριληφθούν, κατά. Ποιο είναι υπέρ του να συμπεριληφθούν αυτέ οι δύο οι λέξει. Να σηκώσει το χέρι του παρακαλώ. Κατά. Α το ελέγξουμε παρακαλώ. Να ψηφίσουμε τι δύο λέξει Labor intensive. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία. να ψηφίζουν μόνο οι... τα μέλη της έκονος τώρα, σας παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Ε, άρα αφαιρούνται οι δύο λέξεις αυτές και τώρα περνάμε στην 33. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την τροπολογία 34. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρασα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική D. Χωρίς προφορική τροπολογία η ψηφορία κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 έως 54. Το ίδιο θέμα έχουν όλες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας αλλάξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά τι γίνεται για την 50 έως και 54. Έναρξη ψηφοφορίας. Τροπολογία διαγραφής. Περισσεύει μια ψήφος από το ΕΛΚ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται την τροπολογία. Ψηφίζουμε τώρα την 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζητείτε έλεγχος ηλεκτρονικός για την 57. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας παρακαλώ. Εάν ψήφισατε όλοι, περισσεύει μία ψήφος από το ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πολύ ωραία. Και τώρα περνάμε στην 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας αλλάξουμε και αυτή ηλεκτρονικά παρακαλώ την 56. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. όλα καταπίπτουν εκτός από την 59. 59. Α, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε, είναι διατύπωση θέμα. Οι 60 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 60 υπέρ. Κατά. Απόχες.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 κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και θα ήθελα να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Να ελέγξουμε, παρακαλώ τα στοιχεία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται το ψήφισμα να ψηφίσουμε τώρα παρακαλώ. Και τώρα εν συντομία παρακαλώ να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει νομοτάτηση της ΕΚΟΝ για να το μεταφράσω σε απλούς όρους. Να ψηφίσουμε και γρήγορα γρήγορα την ε, έκθεση Μπαγιέ. Μία μόνο ψηφοφορία έχουμε. σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 23 του 2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Ποιος είναι υπέρ της γνωμοδότησης αυτής. Να σηκώσει το χέρι του. Και αυτό ηλεκτρονικά. Α, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρα. Η σύσταση εγκρίνεται με 51 ψήφου υπέρ 0 ψήφου κατά και έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίαση της ΕΚΟΝ.